Μπορείτε να καθίσετε κυρίες και κύριοι γιατί πρέπει να ξεκινήσουμε τη συνεδρίασή μας. Έχουμε πολλούς εμπειρογνώμενες από τους οποίους πρέπει να λάβουμε τα φώτα τους και χρειαζόμαστε να έχουμε και χρόνο συζήτησης μεταξύ των μελών και των εμπειρογνωμόνων στη συνέχεια. Να σας ευχηθώ ένα πολύ καλό απόγευμα. Καλώς ήλθατε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, διότι το λέω αυτό στους επισκέπτες αλλά και τις επισκέπτριες. Και ξέρω ότι είναι περιορισμένος ο αριθμός των θέσεων. Δυστυχώς δεν μπορούσαμε να βρούμε πιο μεγάλη αίθουσα συνεδριάσεων, αλλά θα είναι και άνθρωποι που παρακολουθούν στην ε, πρόσθετη αίθουσα παρακολουθήσεως στο 3G2 και έχουμε και το επιγραμμικό μας ακροατήριο στο διαδίκτυο που όλο και αυξάνεται οι εμπειρογνώμονε θα πρέπει να ξέρουν ότι οι ομιλίε του θα καταγραφούν στι ανάδελτου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σε παρεντοσκόπηση τουλάχιστον. Αν έχετε κάτι λοιπόν το οποίο σα ξέφυγε και θέλετε να επανέλθετε, θα υπάρχει πάντα αυτή η δυνατότητα και επίση θα δοθούν και αντίγραφα των διαφανειών στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Δεν ξέρω αν η τεχνολογία μα έχει φτάσει σε σημείο που να μπορεί να βλέπει το ακροατήριο του διαδίκτυου και της διαφάνειας, αλλιώς πρέπει να, τις κατεβα... να τα κατεβάσετε από το διαδίκτυο. Θέλω επίσης να σας πω ότι έχουμε το έγκυρο δελτίο της Επιτροπής μας. Μπορείτε στο πίσω μέρος της αίθουσας να πάρετε αντίγραφα, αλλά μπορείτε και από το διαδίκτυο να δώσετε το ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο και να παίρνετε τακτικά αυτό το δελτίο, το οποίο έχει ηλεκτρονικούς συνδέσμους σε διάφορα έγγραφα. Αυτά υπό παρουσιάσεως. Θα ήθελα λοιπόν να καλωσορίσω τους οκτώ εμπειρογνώμονες στους οποίους θα δώσω διαδοχικό το λόγο και ιδίως θέλω να χαιρετήσω τον Μάρκ Ταραμπέλα, ο οποίος είναι ο εισηγητής της Επιτροπής μας για τις λεγόμενες κλασικές οδηγίες που αρχίζει τώρα να ακούγεται παλιωμοδίτικα αλλά κάποτε θα γίνουν οι σύγχρονες οδηγίες οδηγία για τις κοινοφελείς επιχειρήσεις είναι μία από τις δύο ακροάσεις μας αυτή τη βδομάδα γιατί βλέπω και τον Φιλίπ Ζουβέν που είναι εδώ και είναι ο εισηγητής μας για τις συμβάσεις εκχώρησης, παραχώρησης μάλλον. Οι ρέκτες λοιπόν των συμβάσεων μπορούν να έρθουν και αύριο το πρωί στις 9 να ακούσουν για τις συμβάσεις παραχωρήσεως. Ο στόχος αυτών των ακροάσεων είναι να φέρουμε όσο το δυνατόν περισσότερους εμπλεκόμενους που ενδιαφέρονται για τα θέματα αυτά μαζί μας, να συζητήσουν το σχέδιο μεταρρύθμισης, να μας δώσουν τις απόψεις τους από διαφορετικές οπτικές γωνίες, να ανταλλάξουν απόψεις και με τα μέλη της Επιτροπής μας και να μας βοηθήσουν ούτως εμάς και ιδίω τον εισηγητή στο να απαντήσει στην πρόταση της Κομισιόν. Θα ήθελα στο πλαίσιο αυτό να σας υπενθυμίσω ότι η έχει, η Επιτροπή μας έχει χρειαστεί δυόμιση χρόνια για να προετοιμάσει αυτή τη στιγμή, γιατί <clears throat> εξετάσαμε το πώς λειτουργούν δημόσιες προμήθειες στα κράτη-μέλη. Η κυρία Χάιντι Ρούλε έχει συμβάλει πάρα πολύ από την ομάδα των Πρασίνων και ήταν συγγήτρια δύο εκθέσεων πρωτοβουλία. Κάναμε ήδη μια δημόσια κρόαση, την οποία ήταν πολλοί από εσά. Είχαμε συναντήσει και με εθνικού κοινοβουλευτικού. Είμαστε λοιπόν πολύ καλά προετοιμασμένοι. Μπορούμε να πούμε ότι έχουμε επηρεάσει πολλέ πτυχέ τη μεταρρύθμιση χάρη στι δραστηριότητέ μα. Και αυτό ήταν κάτι που ήταν πολύ σημαντικό τμήμα της εργασίας της Επιτροπής μας. Θέλω ιδιαίτερα να ευχαριστήσω όλες τις πολιτικές ομάδες οι οποίες συμφώνησαν να εργαστούν για ένα θέμα το οποίο mm-hmm. είναι κατά κάποιο τρόπο υπόδειγμα συνεργασίας των Επιτροπών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ήθελα λοιπόν απλώς να, να σας θέσω στο σωστό πλαίσιο. Σε δύο τμήματα θα γίνει η ακρόασή μας τώρα. Καταρχήν θα εστιάσουμε στις στρατηγικές διαστάσεις ε, των δημοσίων συμβάσεων έχοντας σαν κριτήρια την πλευρά του περιβάλλοντος και την κοινωνική πλευρά. Φυσικά μπορούμε εμείς να ετοιμάσουμε το νομοθετικό έργο, αλλά πρέπει κάποιος να το εφαρμόσει επιτοπίως. Και επίσης το θέμα της ισορροπίας μεταξύ ευκαμψίας και ασφάλειας δικαίου. Αυτά είναι τα δύο θέματα τα οποία έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Για κάθε θέμα έχουμε τέσσερις ομιλητές, θα τους παρουσιάσω στη συνέχεια. Θα πρέπει να έχετε τώρα τα βιογραφικά σας, βιογραφικά τους, συγγνώμη, στον φάκελό σας. Οπότε δεν πρόκειται να μπω σε λεπτομέρειες. Απλώς θα τους ζητήσω να λάβουν το λόγο. Θα δώσω λοιπόν στον Μαρκ Τάμπελα το λόγο να κάνει κάποια εισαγωγικά σχόλια για να ενισχύσει και το πλαίσιο που έχω διαγράψει για τη σημερινή ακρόαση. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές. Είναι μεγάλη μου τιμή που βρίσκομαι εδώ δυστυχώς μακριά από τον πρόεδρο. Είναι για να βλέπετε καλύτερα τις διαφάνειες. Όλοι γνωρίζετε ότι το θέμα είναι πολύ σημαντικό γιατί είναι μία, ένα από τα 12 μέτρα που ανακοίνωσε ο Επίτροπος Μπαρνιέ για να καταστεί η εσωτερική αγορά πιο αποτελεσματική. Οι δημόσιες προμήθειες αντιμετωπίζουν πολλές προκλήσεις και τώρα πια έχουμε και κάποια εμπειρία, εγώ έχω δηλαδή, ως τοπικός όπως ήμουν παλαιότερα εκπρόσωπος και έχω κάνει πολλές προσπάθειες να απλοποιήσω τα πράγματα για τους πολίτες και για τις επιχειρήσεις και αυτό πολύ σημαντικό. Γιατί γίνεται πολλής λόγος για την αναθέρμανση της οικονομίας και σε περιόδους κρίσεως όπως αυτή που ζούμε 19% του ΑΕΠ της Ένωσης τι κάνει οφείλεται στις υπηρεσίες. Βέβαια η αλλαγή των κανόνων πάντοτε δημιουργεί και κάποια ανασφάλεια. Εξάλλου δεν έχει μεταφερθεί στην εθνική νομοθεσία το σύνολο των ενωσιακών μέτρων και γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε να μην ξαστοχήσουμε. Ο στόχος, επαναλαμβάνω, είναι η απλοποίηση όλων των διαδικασιών, αλλά και η μεγαλύτερη τους αποτελεσματικότητα για να αντιμετωπίσουν καταλήλως τα προβλήματα που θέτει η ίδια η κοινωνία. Τα προκαταρκτικά τα έχω πει σε ένα έγγραφο εργασίας που κατέθεσα πριν από τρεις εβδομάδες Τα περιβαλλοντολογικά κριτήρια αναφέρονται από την ίδια την οδηγία Πρέπει βέβαια να ξεπεραστούν όλα αυτά γιατί οι εμπειρογνώμονες που ήρθαν σήμερα είναι άνθρωποι που τους έχω συναντήσει πολλές φορές. Εμείς θέλουμε να συναντήσουμε όλους τους ενδιαφερομένους και ενδιαφερόμενες. Είναι πολύ ενδιαφέρον να συναντούμε εκπροσώπους των ενδιαφερομένων γιατί έτσι δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στο πρόβλημά μας και στο πρόβλημά τους. Το πρόγραμμα, το σχέδιο της Επιτροπής που λάβαμε πριν τα Χριστούγεννα δεν είναι ιδιαίτερα ανισχυτικό, αποτελεί μια πρόοδο και το χαιρέτησαν όλοι. Αλλά παρόλα αυτά είναι πολύ πλοκό έγγραφο και πολύ μακροσκελέστερο από μια τρέχουσα οδηγία. Πρέπει λοιπόν να το εξετάσουμε προσεκτικά και σε μερικά σημεία να ενδυναμώσουμε αυτά που λέει, σε άλλα δεν να διορθώσουμε κανονικά. Υπάρχουν και ορισμένες καινοτομίες όπως Euh, Όπως η προβλεπόμενη νέα αυτή εθνική αρχή, και το ενδιαφέρον μιας τέτοιας ακρόασης είναι ακριβώς να ακούσουμε ακόμη και αντιμαχόμενες, αντικρουόμενες απόψεις. Γι' αυτό σταματάω εδώ την εισηγησή μου και θα κάνω μόνο στο τέλος θα βγάλω μερικά συμπεράσματα γιατί σήμερα αυτό που θέλουμε είναι κυρίως να ακούσουμε τους παράγοντες του τομέα αυτού και των επιχειρήσεων, ιδίως των μικρομεσαίων διάφτων, που θέλουμε να λειτουργούν ακόμη πιο αποτελεσματικά, αλλά και τους εκπροσώπους νομικών αρχών, γιατί θέλουμε και απλοποίηση και ισορροπία. Τα νέα κριτήρια να δίνουν τόπο στην καινοτομία αλλά και στη νομική ασφάλεια για να μην δημιουργήσουμε με τα νέα μέτρα ακόμη μεγαλύτερη ανασφάλεια και άρα ακόμη λιγότερη αποτελεσματικότητα. Πρέπει να προσπαθήσουμε λοιπόν να τα βελτιώσουμε όλα. Αυτός είναι τουλάχιστον ο σκοπός μας. Σας ευχαριστώ των προτέρων όλους όσους θα λάβουν το λόγο που θα μας φωτίσουν για το θέμα αυτό που όλοι ξέρουν πόσο πολύπλοκο είναι. Ευχαριστώ Μάρκο για τον ηγετικό σου ρόλο που έπαιξες με τόση ενεργητικότητα. Λοιπόν, ο κάθε ομιλητής 10 λεπτά με το ρολόι. να τηρήσουν αυστηρά αυτόν τον χρόνο ομιλία για να μπορέσει να υπάρξει χρόνος για έρωτα απαντήσεις. Ο δόκτωρ Σάντουιτς Αλμπάνο λοιπόν πρώτος που είναι εκπρόσωπος του Ιταλικού Οργανισμού Προμηθειών. με τίτλο «Αλλαγή στόχων» κλπ έχει πολύ μεγάλη εμπειρία και έχει ασχοληθεί με την κατάστρωση της στρατηγικής της υπηρεσίας του. Με μεγάλη χαρά σου δίνω το λόγο. Με ακούτε? Ναι. Πολύ ωραία. Είναι μεγάλο προνόμιο να βρίσκομαι σήμερα εδώ. Όπως ακούσατε, εργάζομαι για την υπηρεσία CONSIP, την Ιταλική υπηρεσία για τους δημόσιες συμβάσεις. Η εταιρεία μας είναι μια εταιρεία που δημιουργήθηκε πριν από 15 χρόνια και ανήκει στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών με στόχο να εξυγχρονίσει την Ιταλική κρατική διοίκηση. Βασικό τομέα δράση μα είναι η υλοποίηση του προγράμματο για τον εξορθολογισμό των δημοσίων δαπανών για τα αγαθά και τι υπηρεσίε. Και αυτό είναι και ο κύριο λόγο που βρίσκομαι σήμερα εδώ μαζί σα. Η Conship συστηματικά διαδραματίζει σοβαρό ρόλο στο όλο αρχιτεκτόνημα της, ε, του Ιταλικού συστήματος δημοσίων συμβάσεων. Οι όροι μας είναι δεσμευτικοί για την κεντρική κυβέρνηση και εθελούσιας εφαρμογής από τις τοπικές κυβερνήσεις. Όμω επηρεάζουμε τη συμπεριφορά των φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης καθότι πρέπει να ε, καλύπτουν τα κριτήρια ποιότητα τα οποία θέτουμε εμεί με το δικό μα benchmarking. Μα έχει ανατεθεί η αποστολή να ε, δημιουργήσουμε ένα σύνολο κριτηρίων ανάλογα με τις ανάγκες που υπάρχουν δημοσίως και φάνηκε ότι οι δημόσιες συμβάσεις γίνονταν ένα θέμα όλο ένα και πιο περίπλοκο. Υπήρχε λοιπόν η ανάγκη να προσαρμόσουμε την τεχνογνωσία μας για να δούμε πώς μπορούν να οργανωθούν οι δημόσιες συμβάσεις. Υπάρχουν πολλές διαστάσεις που εμφανίζονται και χρειάζεται να εξατεστούν οικονομικά αυτά όμω δεν περιλαμβάνονται στην πρωτογενή και δευτερογενή νομοθεσία κάποια στοιχεία των ε, δημόσιων συμβάσεων, πώς πρέπει αυτά να καταρτιστούν, πώς να οριστούν ε, οι όροι ανάθεσης, πώς να μην υπάρξει σύγκρουση μεταξύ των συμμετεχόντων αλλά και υγιής ανταγωνισμός. Αυτά είναι θέματα που τα έχουμε αναλάβει εμείς και προσπαθούμε να ενημερώνουμε τους ενδιαφερομένους λόγου χάρη για το πρόγραμμα ανταλλαγή δικαιωμάτων εκπομπών. Προσπαθούμε να ευαισθητοποιήσουμε ως προς τους οικονομικούς φορείς τον τομέα <coughs> των πληροφοριών που διαθέτουν για τις διαδικασίες των ε, δημοσίων διαγωνισμών. Αυτό έχει ήδη συμβεί, εφόσον πρόσφατα αναλάβαμε μια συγκεκριμένη προσέγγιση για τον εξυγχρονισμό του συστήματος. Επιδιώκουμε όλο ένα και ευρύτερου στόχους. Το σύστημα των δημοσίων συμβάσεων βασιζόταν σε αυστηρότατες επιλογές, τη χαμηλότερη τιμή ως κριτήριο, ενώ τώρα έχουμε ένα πολύ πιο ευρύ πλαίσιο εξετάζουμε διαφορετικέ δυνατότητε τα επίπεδα ποιότητα, τι οικονομικέ προσφορέ βεβαίω. Αλλά παρόλα αυτά, βασική πρόκληση και θα έλεγα πηγή έμπνευση είναι πώ θα περάσουμε από το αξία για το χρήμα στην κοινωνική αξία για χρήμα. Εδώ υπάρχουν τουλάχιστον τρεις επιπλέον πυλώνες που γίνονται ολοένα θέματα που ευαισθητοποιούν και τους πολίτες. Η βιωσιμότητα, η τοπική διακυβέρνηση και η καινοτομία. Εδώ σημαίνει ότι διευρύνουμε το πεδίο ευκαιριών μπροστά μας, αλλά πρέπει να λάβουμε υπόψη και την περιπλοκότητα του καθήκοντος πρέπει να φέρουμε εις πέρας. Ένα από αυτά τα βασικά καθήκοντα είναι ότι αν θέλουμε να λαμβάνουμε υπόψη περισσότερους συμμετέχοντες στο σχεδιασμό των δημοσίων διαγωνισμών με την κοινωνική πρόνοια λόγω χάρη όπου, αντί, με τον, αντί το κατασκευαστικό τομέα θα πρέπει να δούμε και άλλες πτυχές εξωτερικές δηλαδή περιβαλλοντικές κοινωνικής πρόνοιας Υπάρχει μεγαλύτερο στοιχείο υποκειμενικότητας εδώ. Όταν μιλάμε για περιβαλλοντικές λοιπόν πτυχές στις δημόσιες συμβάσεις, συχνά συμβαίνει το εξής. Δύσκολα διακρίνουμε κάποια ωφέλη από τα κοινωνικά, όμως πρέπει κανείς να τα δει στα πλαίσια ενός ευρύτερου κύκλου, μακρόπνοα, και αυτό πρέπει να κατευθύνει και τη συλλογιστική των δημοσίων δαπανών. Μια άλλη πηγή έμπνευση είναι ότι υπάρχει αποκέντρωση και κάποια φορέ κατακαιρματισμό στι δημόσιε συμβάσει. Δύσκολα λοιπόν οι μικροί συμμετέχοντε μπορούν να επιμείνουν στα κοινωνικά ωφέλη, διότι ενδεχομένω να διαδραματίζουν πολύ μικρό ρόλο σε σχέση με τι μεγαλύτερε, τι γενικότερε δαπάνε. Να λοιπόν πώ αυξάνονται οι πιέσει όταν λαμβάνουμε υπόψη και την κοινωνική διάσταση. Οι κοινωνικές πτυχές γίνονται υποκειμενικότερες, όχι γιατί δεν είμαστε σε θέση να τα κρίνουμε, έχουμε κρίση, αλλά γιατί είναι έργο της κάθε αρχής ανάθεσης να σταθμίσει διαφορετικά το καθένα από τα στοιχεία. Και αυτό είναι ένα από τα ζητήματα που θα πρέπει να το δούμε με εξαιρετική προσοχή και ευαισθησία. Μπορεί εδώ να ανοίξουμε την πόρτα σε πρακτικές διακριτικής μεταχείρισης. Υπάρχει αυτός ο πειρασμός. Μπορεί να υπάρχουν αμφιβολίες για το δίκαιο χαρακτήρα της όλης διαδικασίας του διαγωνισμού. Μπορεί λοιπόν να δοθεί εντύπωση ότι υπάρχουν προκαταλήψεις για μεγαλύτερες κατά μεγαλύτερων εταιρείων μάλλον που δεν είναι τοπικές. Αυτό δεν είναι σύμφωνο με τον σκοπό που έχουμε να δημιουργήσουμε μια ενιαία αγορά προφανώς. Η καινοτομία είναι ένας άλλος πυλώνας και εδώ οι προκλήσεις είναι διτές. Δηλαδή για να μπορέσουμε να πραγματοποιήσουμε καινοτομία πρέπει να αναλάβουμε κινδύνους και οι κρατικοί ε, συμμετέχοντες, μάλλον οι δημόσιοι συμμετέχοντες δύσκολα να λαμβάνουν κινδύνους. Θα πρέπει λοιπόν να αναζητήσουμε τους κατάλληλους διαγωνιζόμενους και να έχουμε την απαραίτητη διαλλακτικότητα και ευελιξία για να πετύχουμε το στόχο μας. Εδώ πρέπει να γίνεται εξάντε από αξιολόγηση της διαδικασίας των δημοσίων ε, προμηθειών κάτι που ε, αυτό καθευτό είναι πολύ καινοτόμο σε σχέση με την ex post ανάλυση, ή ο ανταγωνισμός μάλλον. Τι ρόλο μπορεί να παίξει ως εργαλείο για να επιδιώξουμε και να πετύχουμε τους στόχους μας. Ο ανταγωνισμός είναι κάτι που πρέπει να το δούμε με μία νέα πρόπτικη, ως ένα εργαλείο για να πετύχουμε τους στόχους μας και όχι ως αυτό σκοπό. Όπως θα σας έλεγε κάθε συνετός οικονομολόγος, ο ανταγωνισμός της δημόσιας προμήθειας είναι ένα σημείο πολύ ευαίσθητο, διότι οι δημόσιες συμβάσεις είναι μια διαδικασία που επαναλαμβάνεται συστηματικά. Αλλά αν περιορίσουμε τον ανταγωνισμό σε ένα τέτοιο βαχυπρόθεσμο πλαίσιο, αυτό μπορεί να είναι επικίνδυνο. Θα πρέπει η βάση παροχής να μένει άθικτη μέσα στον χρόνο. Πρέπει να βεβαιωθούμε ότι οι προσφέροντες μπορούν να είναι διαθέσιμοι και αύριο και μεθαύριο και στο μέλλον να κάνουν προτάσεις και να μπορούν να έχουν εμπιστοσύνη στη διαδικασία, στη διαδικασία που θα είναι δίκαιη, που θα βασίζεται σε αντικειμενικά κριτήρια ή τουλάχιστον όσο το δυνατόν αντικειμενικότερα. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι ο ανταγωνισμός πραγματικά στη στιγμή, τη στιγμή της ανάθεσης λαμβάνεται υπόψη Μπορεί λοιπόν έτσι να ε, γίνει ένα εργαλείο στα χέρια μας και να πετύχουμε τις υποσχέσεις που αναλαμβάνουμε σε αυτή τη χρονική στιγμή. Για να υπάρχει ένα δίκαιο λοιπόν επίπεδο ανταγωνισμού πρέπει να ικανοποιηθούν όλες αυτές οι συνιστώσεις ταυτόχρονα. Εάν μπορώ να καταλήξω σε κάποια, δεν θέλω να τα πω συμπεράσματα, θα ήταν ε, ιδιαίτερα ε, υπεροπτικό να το πω αυτό μετά από 10 λεπτά παρουσίασης, αλλά τέλος πάντων κάποιες καταληκτικέ παρατηρήσεις. Οι δημόσιες προμήθειες πρέπει να μπουν σε ένα ρυθμιστικό πλαίσιο, αλλά εύκαμπτο. Όχι με άσκηση διακριτική μεταχείρισης. Επίση, θέλουμε να ενισχύσουμε το σύνδεσμο μεταξύ της κατάρτιση πολιτικών και τι καθημερινέ μα εμπειρίε. διότι η ευρύτερη επιλογή για τους ε, αγοραστές σημαίνει και περισσότερη καθοδήγηση ώστε να μεταφραστούν τα πρότυπα σε καθημερινή πρακτική. Κατά τρίτον, πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι το επάγγελμα των δημόσιων συμβάσεων γίνεται όλο και πιο περίπλοκο. Το προφίλ των απασχολούμενων πρέπει να αλλάξει και επίσης θα πρέπει οι αγοραστές να καταλάβουν ότι η δουλειά τους γίνεται όλο και περισσότερο ρηψοκίνδυνη. Και τέλος, θα πρέπει να δούμε τα θέματα αυτά με μια προοπτική μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Σε 10 χρόνια από σήμερα, να τα ξανασυζητούσαμε, θα βλέπαμε ότι πολλά απομένουν να γίνουν και μερικά δεν τα έχουμε σκεφτεί καν. Θα χρειαστεί λοιπόν να εντείνουμε τι προσπάθειέ μα και να έχουμε υπόψη μας δείκτες για να καταμετρώμε σωστά τα αποτελέσματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο σας ευχαριστώ λοιπόν για αυτά που είπατε και για τους δείκτες που δείξατε για τους επόμενους ομιλητές οι οποίοι θα πρέπει να τα λάβουν υπόψη. Αναφερθήκατε στο θέμα της βιωσιμότητας και για τις πράσινες ε, συμβάσεις. Η Dr. Janet ε, Pritchard, Meissner Pritchard, που είναι επικεφαλής του προγράμματος για τα κλιματική αλλαγή και τα δάση του Client Earth. Έχει δημοσιεύσει ιδιαίτερα στα θέματα αυτά. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας, να μας πείτε τι πιστεύετε για αυτή την πρόταση από την οπτική γωνία της βιώσιμης διαδικασίας ε, συμβάσεων. Έχετε το λόγο για 10 λεπτά. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε. Συγγνώμη, συγγνώμη. Είμαστε μία ΜΚΟ στον τομέα του περιβάλλοντος και ξεκινώντας την παρουσίασή μου θα ήθελα απλώ να σταθώ στους κύριους στόχους που περιέχονται στην έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την οδηγία σε σχέση με τις δημόσιες συμβάσεις, τουλάχιστον αυτούς που γνωρίζω εγώ. Καταρχήν η βιωσιμότητα, η αηφορία, η σαφήνεια, η απλοποίηση και η επίτευξη προσθέμενης αξίας για τους πολίτες. Κατά τη δική μου άποψη, πολλοί από αυτούς οι οποίοι θέλουν να εξασφαλίσουν μεγαλύτερη βιωσιμότητα των ε, ε, συμβάσεων, των δημοσίων συμβάσεων, που είναι και ο λόγος για τον οποίο εμπλεκόμαστε κι εμείς, βλέπουν πολλές φορές ότι αυτοί οι στόχοι βρίσκονται σε ένταση μεταξύ τους, αν όχι σε μετοπική σύγκρουση μερικές φορές. Εγώ όμως θέλω να δείξω με την παρουσίασή μου ότι είναι απαραίτητο, αλλά και εφικτό, να προχωρήσουν χέρι, χέρι αυτές οι οι προτεραιότητες αυτοί οι στόχοι και είναι απόλυτο να συμβαδίζουν αυτοί οι στόχοι για να μπορέσουν να λειτουργήσουν καλύτερα οι πολιτικές στον τομέα των συμβάσεων. Αυτό λοιπόν που εγώ επιδιώκω ως ε, δικηγόρος είναι να υπάρξει πραγματική απλοποίηση και σαφήνεια για να μπορέσει να λειτουργήσει καλύτερα το σύστημα αυτό στην πράξη. Παρά το γεγονό ότι και εμένα με ενδιαφέρει η μεγαλύτερη βιωσιμότητα και είμαι σίγουρη ότι η βιωσιμότητα θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη προσθέμενη αξία. Μέσα στα πλαίσια λοιπόν τη μεταρρύθμιση και τη εξέταση τη πρόταση Κομισιόν θα μπορούσε κανεί να δει ποιε είναι οι κατάλληλε τροπολογίε. Πιστεύω για να το πετύχουμε αυτό θα πρέπει να δούμε καταρχήν ποιε είναι οι βασικέ αρχέ που οι κανόνε για τι δημόσιε συμβάσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθούν να θεσπίσουν Δεύτερον, να συγκρίνουμε τις προτάσεις έναντι αυτών των αρχών και επίσης να προσπαθήσουμε να πετύχουμε ασφ... Ε, σαφήνεια και απλότητα και όχι να μπούμε σε υπερβολική λεπτομέρεια, σε εξαιρέσεις, σε παραδείγματα. Όλα αυτά γίνονται πολλές φορές καλή την πίστη για να επιτύχουμε μεγαλύτερη σαφήνεια, τελικά όμως οδηγούν σε μεγαλύτερη σύγχυση και όχι σε σαφήνεια. Ποιες είναι, ποιες είναι λοιπόν για μένα οι κύριες αρχές σε σχέση με τις δημόσιες προμήθειες και συμβάσεις. Καταρχήν, οι κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι για το πώς γίνεται μία σύμβαση και όχι τι είναι το αντικείμενο της σύμβασης. Πρόκειται για κρατικές αρχές που αγοράζουν πράγματα που χρειάζονται. Αυτές οι αρχές πρέπει να αγοράσουν λοιπόν αυτό το οποίο θέλουν και πρέπει να καθορίσουν οι ίδιες τι είναι αυτό το οποίο επιζητούν να αγοράσουν. Μια δεύτερη βασική αρχή, ιδίω σε ό,τι αφορά τη βιωσιμότητα, είναι ότι θα πρέπει <clears throat> οι οριζόντιοι επιζητουν να αγορασουν μια δευτερη βασικη αρχη ιδιως σε οτι αφορα τη βιωσιμοτητα ειναι οτι θα πρεπει οι οριζοντιοι στοχοι να έχουν την ίδια αξία με τους λειτουργικούς στόχους. Για μένα αυτό σημαίνει ότι έχουμε διπλή αγοραστική δύναμη για τις συμβάσεις. Αν λοιπόν μια αρχή θέλει να αγοράσει ανακυκλωμένο χαρτί και όχι απλώς χαρτί, δεν αγοράζει μονάχα ε, το χαρτί αυτό, αλλά αγοράζει και μία αποδοτικότητα στη χρήση των υλικών πόρων. Γι' αυτό λέω ότι είναι μία διπλή μορφή αγοράς. Υπάρχουν λοιπόν περιπτώσεις που ισχύει αυτό μέσα στα πλαίσια του υποθέσεων που έφτασαν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, που τόνισε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ότι οι οριζόντιοι στόχοι είναι ίσης αξία με τους λειτουργικού στόχους και έχουν εφαρμόσει μια διασταλτική εμπειρία για το τι σημαίνουν αυτοί οι οριζόντιοι στόχοι. Μια τρίτη σημαντική αρχή είναι η καλύτερη αξία σε σχέση με το κόστος. Επανέρχομαι σε αυτά που είπα, νομίζω ότι είναι σαφές ότι το να έχουμε πιο βιώσιμη και αηφόρο διαδικασία δημοσίων συμβάσεων δίνει την καλύτερη αξία και την καλύτερη αποτελεσματικότητα στις δαπάνες. Και επίσης σε σχέση με την αηφορία είναι απαραίτητο από τη Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως περιλαμβάνεται στην αρχή της ε, ενσωμάτωσης <clears throat> και υποστηρίζεται με τις αρχές των ε, σχεδίων δράση για βιώσιμη παραγωγή και κατανάλωση. Επομένως, οι δημόσίε αρχέ είναι ένα σημαντικό εργαλείο για να εξάρουμε τις αξίες της βιώσιμη ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μια τέταρτη αρχή είναι η σύνδεση με, τον... <coughs> με το αντικείμενο. Ο κανόνας που λέει ότι πρέπει να είναι συν... που να συνδέεται η σύμβαση με το αντικείμενο. Αυτό μπορεί κανείς να θεωρήσει ότι ορισμένοι λένε ότι είναι υπέρ, αλλά ότι είναι κατά τη βιώσιμότητα. Εγώ πιστεύω ότι αυτό ο κανόνα θα πρέπει να ερμηνευτεί με σωστό τρόπο, γιατί όταν λέμε ότι θέλουμε να επιτύχουμε οριζόντιου στόχου μέσω των συμβάσεων, υπάρχουν ανησυχίε πολλέ φορέ ότι αυτό μπορεί να είναι άνοιγμα των ασκών του αιώλου και μπορεί να επιτρέψει περίπου το οτιδήποτε. Και ότι προσπαθούμε να αλλάξουμε τα πράγματα μέσα από τι δημόσιε συμβάσει και όχι με του καλύ... με με τις κατάλληλες ρυθμιστικές ενέργειες. Η σύνδεση λοιπόν με το αντικείμενο είναι σημαντική αρχή γιατί εμποδίζει μια υπερβολική χρησιμοποίηση των οριζόντιων αρχών πέρα από το συγκεκριμένο θέμα δημόσιας προμήθειας. Και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ήταν πάρα πολύ σαφές σε σχέση με το γεγονός ότι είναι σημαντικός αυτός ο κανόνας, συγχρόνως δίνοντας μια ιδιαίτερα ευρεία ερμηνεία σε σχέση με το τι σημαίνει συνδεόμενο με το αντικείμενο. Τέλος έχουμε τις αρχές της διαφάνειας και ισότητος προστασίας και αυτές είναι σημαντικές αρχές. Θεωρώ ότι αυτές είναι οι κέρυες αρχές οι οποίες εξασφαλίζουν αυτούς οι οποίοι υποβάλλουν προσφορές στη διαδικασία. Κάτι το οποίο μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα μετά από αυτά που είπε και ο προηγούμενος ομιλητής για να εξασφαλίσουμε μια ισοδίκαια μεταχείριση όλων των των προτάσεις, να εξασφαλίσουμε ότι έχουμε την καλύτερη αξία που μπορούμε να αποσπάσουμε από μια τέτοια διαδικασία προσφορών και να εξασφαλίσουμε ότι υπάρχει η συμμεταχείριση και ισότηση ευκαιριών και πέραν των εθνικών συνόρων. Αν λοιπόν ο στόχος μας είναι να επιτύχουμε μια απλοποίηση και μεγαλύτερη σαφήνεια, ώστε να έχουμε μεγαλύτερη βιωσιμότητα και αηφορία στα θέματα αυτά, θα πρέπει <clears throat> να αποφύγουμε την υπερβολική πολυπλοκοποίηση των κανόνων. Για μένα οι κανόνες αυτοί γίνονται πολύπλοκοι όταν δεν σεβόμαστε την αρχή της ισορροπίας και της εμπιστοσύνης όταν μπερδεύουμε τους οριζόντιους στόχους με τους λειτουργικούς στόχους και όταν δεν χρησιμοποιούμε τον κανόνα σχέση με το αντικείμενο για να μην υπάρξει υπερβολική χρήση κάποιων αρχών. Και επίσης υπάρχουν προβλήματα όταν δεν έχουμε τις αρχές της διαφάνειας και της ίσης προστασίας. Και μέσες φορές βασιζόμαστε υπερβολικά στις αρχές αυτές της διαφάνειας και της ισότητας και θεωρούμε ότι αυτές και μόνο θα πρέπει να είναι ο κύριος γνώμονας στις ενέργειες αγοράς. Για να έλθω λοιπόν σε κάποιες συγκεκριμένες ρήτρε της οδηγίας, το άρθρο 40 για παράδειγμα που αφορά στις τεχνικές προδιαγραφές. Στην προτινόμενη μεταρρύθμιση, το άρθρο αυτό ξεκινά λέγοντας ότι οι τεχνικές προδιαγραφές μπορεί να περιλαμβάνουν οριζόντιους στόχους, και ακόμα πιο ειδικά η πρόταση προχωρά και λέει ότι οι διαδικασίες που εμπλέκονται στην παραγωγή και άλλες μη χρηστικές φάσεις του κύκλου ενός εργαλείου μπορούν να επεμβαίνουν στους οριζόντιους στόχους. Αλλά οι λεπτομέρειες του άρθρου 40 στη συνέχεια περιορίζουν τις τεχνικές προδιαγραφές σε επίτευξη λειτουργικών και μόνο στόχων. Υπάρχει λοιπόν έλλειψη συνεκτικότητος στο άρθρο 40 και δεν υπάρχει ασφάλεια δικαίου και σαφήνεια δικαίου. Το ίδιο ισχύει και στο, στο αιτιολογική σκέψη 41 που λέει ότι η σύνδεση με το αντικείμενο είναι βασικό στοιχείο για τις τεχνικές προδιαγραφές και αυτό περιλαμβάνει τις, ε, τον ορισμό των χαρακτηριστικών παραγωγής. Λέει όμως στη συνέχεια -hmm. ότι διάφορε πτυχέ που έχουν να κάνουν με την κοινωνική βιωσιμότητα στην παραγωγή μπορούν να θεωρηθούν ότι είναι κριτήρια απονομή μια σύμβαση και όχι τεχνικέ προδιαγραφέ. Αυτό λοιπόν μπορεί να δημιουργήσει πράγματι σύγχυση όταν πρόκειται για μια αρχή η οποία πρέπει να αποφασίσει σε ποιον θα δώσει μια σύμβαση. Πώ λοιπόν μπορούμε να πετύχουμε να έχουμε μια σαφήνεια σε σχέση με τα θέματα αυτά και τη διαδικασία ε, προμηθειών και τις τεχνικές προδιαγραφές πιστεύουμε ότι αυτά τα οποία θα πρέπει να θεωρούνται ως τεχνικές προδιαγραφές έναντι των κριτηρίων απονομής θα πρέπει να βασίζονται στην έννοια του, της σύνδεσης με το αντικείμενο ευρεία τη έννοια. Η διαφορά μεταξύ των δύο δεν έχει να κάνει με την ουσία των κριτηρίων, δηλαδή το αν έχουν να κάνουν με παραγωγή, με χρήση ή αν συμβάλλουν στους οριζόντιους λειτουργικούς στόχους ή αν έχουν να κάνουν με την κοινωνική αηφορία ή την περιβαλλοντική αηφορία. Αντίθετα, η διαφορά μεταξύ των τεχνικών προδιαγραφών και των κριτήριων απονομή μια σύμβαση έχουν να κάνουν με τη λειτουργία των δύο αυτών στην διαδικασία λήψη αποφάσεων για τη σύμβαση. Έχουμε λοιπόν δύο διαφορετικά εργαλεία τα οποία επιτρέπουν την αρχή που διενεργεί ένα διαγωνισμό να αποφασίσει τι θέλει να αγοράσει και να έχει τη σωστή πληροφορία στην κατάλληλη στιγμή για να κάνει την καλύτερη απόφαση σε σχέση με την επιδιωκόμενη αξία. Οι τεχνικές προδιαγραφές πρέπει να είναι απόλυτες αναγκαιότητες από την πλευρά της αρχής του διαγωνισμού. Αν δεν μπορούν λοιπόν οι υποβολές προτάσεων να ικανοποιήσουν τις τεχνικές προδιαγραφές, δεν μπορούν να συμβάλλουν, δεν μπορούν να ανταγωνίζονται για την σύμβαση αυτή. Αν πει κανείς παραδείγματος χάρη ότι θα αγοράσει μονάχα ηλεκτρισμό από ανανεώσιμες πηγές, μπορούν να το πράξουν αυτό μπορούν να πούνε ότι αυτό είναι τόσο σημαντικό παραγωγός χάρη να ενισχύσουν θέματα κλιματικής αλλαγής που χρησιμοποιούν μόνο αυτό το κριτήριο. Αντίθετα, τα κριτήρια απονομής μιας σύμβασης επιτρέπουν στην αρχή να εξισορροπήσει διάφορες αξίες μεταξύ τους. Ο καθένας κάνει κάθε μέρα τις επιλογές του σε σχέση με την αγορά ενός προϊόντος. Το κάνουμε όλοι σε επίπεδο καταναλωτών. Για το ίδιο παράδειγμα, μπορεί να παίρνει μια υποβολή πρότασης πρόσθετα μόρια αν ενισχύει την ανανεώσιμη ενέργεια, αλλά και αυτό πρέπει να εξορροπηθεί έναντι της τιμής ε, παροχής ηλεκτρισμού. Πρέπει λοιπόν να δούμε το πώς κάθε λεπτομέρεια μέσα σε μια υποβολή, μέσα σε μια προκήρυξη σύμβασης ανταποκρίνεται στις βασικές αυτές αρχές. Εάν δεν διευκρινίζει και δεν ικανοποιεί τις βασικές αυτές ε, αρχές, δεν έχει νόημα η οδηγία να είναι αυτό το οποίο δεσμεύει τις αρχές του, των συμβάσεων. Δεν, δεν ήμουν αυστηρός με το χρόνο σας. Αλλά υπενθυμίζω στους υπόλοιπους ότι δεν θα είμαι τόσο ανεκτικός. Σας κατευχαριστώ και οι δύο παρουσιάσεις μέχρι τώρα είχαν κοινό θέμα και συμπληρωματικές παρατηρήσεις. Τώρα θα μιλήσει η Βερόνικα Νίλσεν που είναι γραμματεύς για τις δημόσιες προμήθειες στην Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Συναδικάτων έχει μεγάλο παρελθόν στα συνδικάτα και ιδιαίτερα στο θέμα των προμηθειών. Έχει το λόγο για 10 λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πρέπει να σας πω ότι στην Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Συνδικάτων έχουμε μια αναθεωρημένη οδηγία για τις προμήθειες, για το σεβασμό των συνθήκων εργασίας και για την κοινωνική πτυχές, την ποιότητα των υπηρεσιών κλπ. Ξέρω ότι το λάβατε γιατί το είδα εκεί στα χαρτιά. Τώρα όμως θα βασιστώ στα κοινωνικά κριτήρια που είναι διαφορετικό θέμα. Πώς ορίζονται αυτά και κυρίως πώς εφαρμόζονται. Είναι σημαντικό να ξέρουμε ότι δεν μπορούν όλα να λυθούν από τις δημόσιες προμήθειες. Για μας η βασική αρχή είναι η πειθαρχία στις συλλογικέ συμβάσεις και τον εθνικό νόμο για τις προμήθειες. Αυτό μπορεί να σας φαίνεται πολύ απλοϊκό γιατί ο σεβασμός του νόμου είναι κάτι το στοιχειώδες αλλά το θέμα είναι ότι πολλές φορές η εργασιακή νομοθεσία, η εργατική νομοθεσία παραβιάζεται. Στην πρόταση της Κομισιόν η δυνατότητα να συμπεριληφθούν τα κοινωνικά και τα περιβαλλοντολογικά στις προμήθειες είναι, δεν είναι υποχρεωτική για τους συμβαλωμένους. Εμείς δεν συμφωνούμε με αυτό και ζητούμε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να κάνει να τις καταστήσει δεσμευτικές αυτές τις ρήτρες. Η ίση μεταχείριση στον τόπο εργασίας είναι κάτι το πολύ βασικό οι θεσμοί της Ένωσης πρέπει να διασφαλίζουν ότι το πλαίσιο δημοσίων προμηθειών θα σέβεται όλους τους όρους για την απασχόληση στον τόπο της εργασίας και επίσης να διασφαλίζει ότι θα είναι συμβατός ο Ευρωπαϊκός νόμος με τις συνθήκες του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας που προβλέπουν ότι δεν πρέπει καμία διάταξη να είναι πιο απαγορευτική από εκείνη που ισχύει με τις συλλογικές συμβάσεις για το ίδιο θέμα. Πιο συγκεκριμένα οι κανόνες δημοσιοφορμηθειών πρέπει να συμπεριλαμβάνουν την απέτηση να εφαρμόζονται όλες οι διατάξεις του νόμου για την εργασία, του εργατικού νόμου. Όταν βέβαια δεν υπάρχει εποπτεία και υπεργολαβίες είναι δύσκολο να δει κανεί αν γίνονται σεβαστά σε όλες οι διατάξεις του νόμου. Έτσι είναι αδύνατο από τη μία η δημόσια συμβαλόμενη αρχή να ταυτίσει καν πιο σε ευθύνεται ακριβώς για τις παραβιάσεις των συλλογικών συμβάσεων και του εργασιακού νόμου. Γι' αυτό πρέπει να ε, είναι υποχρεωτικό να ισχύουν οι δίτρες αυτές και για τους υπεργολάβους. Νομίζουμε ότι πρέπει να υπάρξει ένα σύστημα σαφούς καθορισμού των ευθυνών ώστε η κοινωνική προστασία, τα βασικά δικαιώματα, η πληρωμή να γίνονται σεβαστά. Οι δημόσιες προμήθειες με βάση το χαμηλότερο κόστος αντιτίθενται συνήθως στην αρχή του σεβασμού των κοινωνικών ρητρών. Βέβαια λόγω της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης και των περικοπών είναι προφανές ότι όλο και περισσότερες αρχές θα δίνουν τα συμβόλαια στον, στον χαμηλότερο, στον μεγαλύτερο μειοδότη. Και αυτό μπορεί να μην συμβαδίζει με το σεβασμό των περιβαλλοντολογικών και εργασιακών ρητρών. Και έτσι μπορεί να χειροτερεύσουν και οι συνθήκες εργασίας και η ποιότητα των προϊόντων. Στη Δανία τα δανεικά συνδικάτα εξέτασαν κατά πόσον υπήρχαν εξοικονομήσεις από τη χορήγηση συμβολέων σε εξωτερικές υπηρεσίες θεωρήθηκε ότι υπήρχε μείωση του κόστους κατά 50% αλλά τα συνδικάτα θεώρησαν ότι οι καινούργιες αυτές εταιρείε χρησιμοποιούσαν προσωπικό με χαμηλότερα προσόντα και δεν πλήρωναν τις υπερορίες. Αλλά στη Δανία βέβαια υπάρχουν και καλές εμπειρίες για τη διασφάλιση του σεβασμού των εργασιακών συνθήκων και των νόμων. Υπάρχουν παραδείγματα από συμβόλαια που χορηγήθηκαν στο Δήμο της Κοπενχάγης που είναι πολύ θετικά, αλλά επειδή υπάρχει και ένας δανός εκπρόσωπος εδώ μπορεί αυτός να τα πει καλύτερα. Άλλο παράδειγμα από τη Γερμανία Υπάρχουν στοιχεία που λένε ότι οι δημόσιες αρχές χορηγούσαν συμβόλαια με την αρχή της μειοδοσίας και αυτό κατέληξε σε μείωση των μισθών και των συνθήκων εργασίας. Αυτό ήταν το πρώτο από τα κριτήρια της Κομισιόν, το χαμηλότερο κόστος. Το δεύτερο είναι το πιο ποιοτικά συμφέρον συμβόλαιο. Ποιότητα αναφέρεται εκεί, αισθητικά και λειτουργικά στοιχεία, περιβαλλοντολογικά και στοιχεία καινοτομία. Δεν υπάρχει όμως τίποτε για τα κοινωνικά, κανένα κοινωνικό κριτήριο. Νομίζουμε λοιπόν ότι η οδηγία πρέπει να προσθέσει κριτήρια. Παραδείγματο χάρη μια τοπική αρχή σε περιοχή υψηλής ανεργίας μπορεί να θέλει να βάλει μια ρήτρα που απαιτεί ε, από ορισμένους άνεργους να χρησιμοποιηθούν για την πραγματοποίηση του συμβολέου. Τέτοιες ρήτρε λοιπόν για τους ανέργους και για τα προσόντα πρέπει να είναι δυνατόν να συμπεριλαμβάνονται σε αυτή την οδηγία. Η κοστολόγηση με βάση όλον τον βιολογικό κύκλο είναι μια άλλη ιδέα. Παραδείγματο χάρη. Στην πρόταση της Κομισιόν δεν αναφέρονται ακόμη μία φορά οι κοινωνικές πτυχές της υπεργολάβησης και υπεργολαβίας. Και αυτά, αυτό κόστος είναι κοινωνικό όμως κόστος. Τα ε, περιέργως, οι περιέργως χαμηλές προσφορές είναι συνήθως εκείνες που οδηγούν στο μεγαλύτερο κοινωνικό ντάμπινγκ. Αν μια προσφορά φαίνεται περιέργως χαμηλή πρέπει να αποδεικνύει ο προσφέρον ότι θα σεβαστεί όλες τις συνθήκες εργασίας που προβλέπονται από τον νόμο. και κατά την εκτέλεση του συμβολέου κάθε παραβίαση των συνθηκών εργασίας πρέπει αυτομάτως να οδηγεί στην κατάργησή του. Η πρόταση της Κομισιόν μιλάει για την δυνατότητα πιστοποιήσεων για την εγγύηση της ε, νόμιμης συμπεριφοράς των συμβαλωμένων ή των προσφερόντων ότι θα σέβονται και το περιβάλλον και τις συνθήκες εργασίας και ε, εγγύηση ότι τα κριτήρια ποιότητας μπορούν να οδηγήσουν σε βελτίωση της ποιότητας του προγράμματος των συνθηκών εργασίας και ακόμη και των μισθών. Επίσης θα ήθελα να τονίσω ότι όπως γνωρίζετε στην οδηγία προβλέπεται ειδικό καθεστώς για τις κοινωνικές υπηρεσίες, πράγμα το οποίο δεχόμαστε, αλλά πιστεύουμε ότι πρέπει να συμφωνεί με τους ισχύοντες εθνικούς νόμους και τις συλλογικέ συμβάσεις. And finally, Τέλος, θα, τελειώσω πριν από τα 10 λεπτά, δεν πειράζει. Υπάρχει ο οδηγός της Κομισιόν από το 2010 για τις κοινωνικές πτυχές των δημοσίων προμηθειών γιατί είναι και αυτό μια βάση ορισμού των κοινωνικών κριτηρίων έχουν ορίσει ορισμένες κατηγορίες συμφωνίας με τους ισχύοντες νόμους για την εργασία και μερικά άλλα κριτήρια τα οποία δεν αναφέρω γιατί τα σημαντικότερα είναι αυτά που σας είπα. Well, Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή την σαφέστατη παρουσίαση. Ακριβώς τα 10 λεπτά φτάσατε. Αλλά ε, ήταν ε, πολύ ευρύ το υλικό που καλύψατε σε μια τόσο σύντομη παρουσίαση. Θα σας θέσουμε ερωτήματα αργότερα. Και τώρα για να ολοκληρώσουμε αυτό το γύρο μιλητών, να καλωσορίσω έναν άλλον εμπειρογνώμονα για τις δημόσιες συμβάσεις από την Δανία που ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή έχει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ακούσαμε τη δέσμευση της Δανέζικης Κυβέρνησης για να αναλάβει πρωτοβουλίες για τις δημόσιες συμβάσεις γενικότερα. Γι' αυτό είναι παρόν και το Συμβούλιο. Ο Γιάκομ Σάρφ έχει μεγάλη πείρα στις δημόσιες συμβάσεις, εργάζεται αυτή τη στιγμή στο Δανικό Εμπορικό Επιμελητήριο, ενώ προηγουμένως ήταν υπεύθυνο του της πύλης για τι δημόσιε συμβάσει τη δανεικής κυβέρνηση. ένα από τα καλύτερα παραδείγματα πρακτικών που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλό θα ήταν να ακολουθήσει στι διατάξει ε, τη σημερινή πρόταση. προκειμένου να βελτιώσει την ποιότητα των δημοσίων συμβάσεων γενικότερα και την συμμόρφωση στα κράτη-μέλη. Θα μα μιλήσει για την προοπτική των επιχειρήσεων και το πώς εργάζεται κανείς με κοινωνικά και πράσινα κριτήρια. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε, αγαπητοί και αγαπητές βουλευτές. Ευχαριστώ για την ευκαιρία να προσέλθω σήμερα για να σας παρουσιάσω τις εμπειρίες μας για το πώς λειτουργούν οι δημόσιες συμβάσεις και ποια είναι η στρατηγική τους χρήση. Θα ακολουθήσω μια διαφορετική σκοπιά από τη Σουηδή, συνάδελφο. Απλώς ορισμένες παρατηρήσεις για να ξεκινήσουμε. Πρώτα απ' όλα, Έρχομαι από μια ένωση επιχειρήσεων. Εκπροσωπούμε 17.000 δανεικές επιχειρήσεις, εκ των οποίων πολλέ και από τον δημόσιο τομέα στη Δανία. Ασχολούνται με τι δημόσιε συμβάσει σε καθημερινή βάση. Στι συνομιλίε μα στη Δανία αυτή τη στιγμή μα ενδιαφέρει κατά πόσον θα μπορούσαμε να είχαμε ένα καλύτερο σύστημα δημοσίων συμβάσεων. Θα ξεκινήσω λοιπόν από την εξή διαπίστωση και νομίζω όλοι μπορούμε να συμφωνήσουμε. Οι μικρομεσαίε επιχειρήσει. και πολλά από τα μέλη τη Ένωσή μα είναι μικρομεσαίε επιχειρήσει, βρίσκονται στην καρδιά τη δημιουργία θέσεων εργασία στην Ευρώπη και γενικότερα τη ε, ανάπτυξη στην Ευρώπη. Αυτό δεν νομίζω ότι χρειάζεται καν να το συζητήσουμε. Έπειτα, όταν μιλάμε για δημόσιε συμβάσει, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι πολύ ευάλωτες στα στις περίπλοκους κανόνες, στα μεγάλα, στο μεγάλο κόστος των συναλλαγών, <clears throat> το άχθος της διεξαγωγής μελετών. Θα μπορούσε μια δανεική εταιρεία να δαπανίσει 31.000 ευρώ για τέτοιου είδους προσφορές, συμμετοχές μέλλον. Εάν αυτά τα μεταφράζαμε σε δανεικέ κορώνες, θα ήταν 4,6 εκατομμύρια. Πάρα πολλά χρήματα σε ευρωπαϊκούς όρου. Και αυτό γιατί οι κανόνε είναι πολύ περίπλοκοι. Όταν συζητά κανεί λοιπόν τις πράσινες ε, συμβάσει τι κοινωνικέ συμβάσει και αυτό μας απασχολεί από τη σκοπιά των μικρομεσών επιχειρήσεων, είναι να καταλήξουμε να πούμε ότι είναι πολύ περίπλοκοι κανόνε. Μεγάλο το άγχο, ιδίω αυτό που επομίζονται οι μικρομεσαίε. Εάν θέλουμε λοιπόν να δημιουργήσουμε περισσότερε θέσει εργασία, δεν είναι αυτό ο σωστό τρόπο να προχωρήσουμε. Δεν πρέπει η νέα πρόταση να έχει περίπλοκου κανόνε. Αν το διαβάσετε, είναι 100 σελίδε χωρί τα παρατήματα. Κάποια από τα μέλη τη Ένωσή μα δεν έχουν καν ε, πτυχία νομική ή νομικές υπηρεσίες για να μπορέσουν να συμμετέχουν για να κάνουν τις προσφορές τους στους οποιοδήποτε, στους οποιοδήποτε διαγωνισμούς μπορεί να προκηρυχθούν. Για το πλαίσιο τώρα, το νομικό πλαίσιο, νομίζουμε ότι ήδη λειτουργεί. Νομίζω θα το σχολιάσω σε λίγο. Το ίδιο και για τις ε, προμήθειες υπηρεσιών. Όταν σταθούμε όμως στο θέμα της καινοτομία, βλέπουμε ότι το σημερινό πλαίσιο αλλά και η πρόταση που σήμερα Μα έχει υποβάλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με κάθε συμβασμό, νομίζουμε ότι είναι άθλια. Εάν μιλήσουμε για πράσινες προμήθειες, νομίζω ότι είναι ευρέω αναγνωρισμένο ότι η Δανία ε, είναι μια από τις πρώτε χώρες που ανέπτυξε τις ε, πράσινες δημόσιες προμήθειε είναι αναπόσπαστο στοιχείο το πράσινο των ε, δημόσιων συμβάσεων στη Δανία και μάλιστα θα προχωρήσουμε κι άλλο. Πώς προοδεύσαμε τόσο. Ακολουθώντας την προσέγγιση κατά πρώτον του να κάνουμε ότι είναι εφικτό. Εφόσον είχαμε τις δυνατότητες σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Αυτή η προσέγγιση λειτουργήσε από κάτω προς τα πάνω και όχι αντίστροφα. Πολλές χώρες Νομίζω θα πρέπει να ακολουθήσουμε αυτό το παράδειγμα όταν μιλάμε για πράσινες προμήθειες. Τι μπορέσαμε να... Τι θέσαμε σε εφαρμογή μάλλον, εταιρικέ σχέσεις μεταξύ κυβερνήσεων, ε, ενώσεων επιχειρήσεων, συμβάλλουσες αρχές, μη κυβερνητικές οργανώσεις, τοπικούς φορείς. Ε, Γενικώ οργανωθήκαμε για να δούμε πώς μπορούμε να σχεδιάσουμε σωστά τις πράσινες δημόσιες συμβάσεις. Και δημιουργήσαμε κατευθυντήρες γραμμές και εργαλεία, μιλήσαμε με τις συμβάλλουσες αρχές, αν δείτε το διάγραμμα στην εικόνα, πέρσι αυτό το consortium, αυτός ο όμιλος για τις πράσινες ε, προμήθειε, ζήτησε από τις συμβάλλουσε αρχέ, τι θα σας έκανε να αγοράσετε περισσότερο πράσινο. Μα είπαν καλύτερες κατευθυντήριες γραμμές, ε, καλύτερη διαχείριση μάλλον και καλύτερη γνώση για το πώ λειτουργούν τα πράσινα προϊόντα. Δεν μα ζήτησαν πρωτογενή νομοθεσία. Δεν είχαμε τέτοια αιτήματα. Ούτε μα είπαν ότι χρειαζόμαστε συγκεκριμένα προγράμματα πράσινων προμηθειών. Όχι, δεν ήταν αυτά τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου μα. Προερχόμενο λοιπόν από μια χώρα που έχει διανύσει πολύ δρόμο, μπορώ να σα πω τι λειτουργήσε για μα και νομίζω και για άλλε χώρε. Να τονίσω ότι ακόμη πολλά μπορούν να γίνουν και ιδίω ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη θα μπορούσαν να αναπτύξουν τέτοια μοντέλα TCO όπως ονομάζονται, ώστε να ληφθεί υπόψη και η οικονομία και η βιωσιμότητα και η καινοτομία. Και μάλιστα θα πρέπει να, είμαστε, να έχουμε δύο μοντέλα για να προχωρήσουν τα πράγματα περισσότερο. Για τι κοινωνικέ τώρα δημόσιε συμβάσει. Εδώ τα πράγματα διαφέρουν αρκετά σε σχέση με τι πράσινε. Πολλέ φορέ έχουμε να κάνουμε με ανέργου, με ανθρώπου με ειδικέ ανάγκε, ανάπηρου, οι οποίοι στους οποίους μάλλον θα ζητηθεί να εργαστούν για κάποια από τα μέλη της Ένωσής μας. Μιλάμε για ανθρώπους με ιδιαίτερες ανάγκες. Πώς θα αντιμετωπίσαμε αυτό στη Δανία και το προωθήσαμε μάλιστα σε ένα βαθμό. Με κοινωνικές εταιρικές σχέσεις και τη χρήση αυτού που ονομάζουμε κοινωνικές ρήτρε στις κοινωνικές συμβάσει. Δεν θεωρούμε ότι είναι η μαγική λύση, ούτε τέλεια συνταγή, αλλά το δοκιμάσαμε, εργαστήκαμε με βάση αυτό το εργαλείο και πάλι από τα κάτω προς τα πάνω. Δηλαδή, Βλέπετε εδώ ε, μια εικόνα από τη διαφημιστική μας εκστατεία του 2001 και πραγματικά όταν πηγαίνει κανείς και μιλά στις συμβάλλουσες αρχές της επιχειρήσης και λέει ότι χρειάζονται ευκαιρίες συμπερίληψης ανέργων, ανθρώπων με δικές ανάγκες μέσω των δημοσίων διαγωνισμών. Κάποιο αποτέλεσμα υπάρχει. όμως πρέπει να πω και το εξή. Α μην απατώμεθα. Όταν ξεκινήσαμε στη Δανία με αυτό το σύστημα, είπαμε Ίσως να μπορέσουμε να βάλουμε από την πίσω πόρτα χιλιάδες και χιλιάδες ε, αναπήρους ε, σε θέσεις εργασίας. Εντάξει, δεν είναι αυτό το αποτέλεσμα, δεν είναι εφικτό για πολλούς διαφορετικούς λόγους. Δεν μπορεί να γίνει αυτό με τις ε, κοινωνικές δημόσιες συμβάσεις. Αυτή είναι η σκληρή πραγματικότητα. Ναι, χρήση των κοινωνικών ρητρών, αλλά όπου είναι και λογικό. Ακόμη λογικότερο είναι να ενσωματώσουμε, μάλλον να συνάψουμε σχέσεις, κοινωνικές εταιρικέ σχέσεις με αρχές από τη μια που εκπροσωπούν ανθρώπου με ειδικέ ανάγκε και ιδιωτικέ επιχειρήσεις από την άλλη. Είδαμε παράδειγμα την περασμένη εβδομάδα από αλυσίδα ε, σούπερ μάρκετ που προσέλαβε ανθρώπου με ειδικέ ανάγκε. Δεν ήταν δημόσιο διαγωνισμός αυτός, ήταν ένας ιδιωτικό ε, επιχειρηματίας που πίστεψε ότι κάνοντας αυτή την κίνηση κάνει κάτι καλό για την επιχείρησή του και για του πολίτε. Και πάλι δεν μιλάμε αναγκαστικά για ρύθμιση σε ευρωπαϊκό όμω επίπεδο. Προχωρούμε τώρα στην καινοτομία. Τι βλέπουμε. Υπάρχουν παραδοσιακοί δημόσιοι διαγωνισμοί, εκατοντάδες, που εντοπίζονται στη χαμηλότερη τιμή. Αυτό δημιουργεί άκαμπτες διαδικασίες, πολύ δεσμευτικέ. Είναι πια η στιγμή να ήρθε καιρό να δημιουργήσουμε ένα περισσότερο ε, εύκαμπτο σύστημα να υπάρχει ε, διάλογο στη διαδικασία τη διαπραγματεύση. Ναι, καινοτόμε εταιρικέ σχέσει, όπω το λέει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά όχι μόνο για ειδικέ περιπτώσει, όπω τώρα το παρουσιάζει το άρθρο 24 τη πρόταση. Βλέπουμε πολλές φορές να υπάρχει ε, κακή διαχείριση, κακοδιαχείριση των δημοσίων κονδυλίων. Γιατί ακριβώς είναι περίπλοκες οι διαδικασίες πρέπει εδώ λίγο να σταθώ και στο σύστημα της Δανίας, το οποίο θεωρείται ένα ήπιο σύστημα δημοσίων συμβάσεων, δεν είναι αυτό που βασίστηκε στις κλασικές οδηγίες, είναι κάτω από το όριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και μιλάμε για τις υπηρεσίες που αναφέρονται στο παράρτημα Β, στις ήπιες υπηρεσίες όπως λέγονται, τις soft services, και ούτω καθεξής. Κάποια κράτη-μέλη το δέχτηκαν αυτό. Υπάρχει λοιπόν και σε άλλες εθνικές νομοθεσίες τέτοιου είδους ρύθμιση. Κάπως έτσι θα είναι το αποτέλεσμα. Τι λέει ακριβώς λοιπόν ο δικός μας ο νόμος. Ότι αν αγοράσει κανείς κάτι πάνω από το όριο των 6.500 ευρώ περίπου, δεν υπάρχουν ε, υποχρεώσει. Βασικέ αρχέ τη συνθήκη, ναι, πρέπει να γίνονται σεβαστέ. Δεν λέμε όμω στι συμβάλλουσε αρχέ ότι πρέπει να χρησιμοποιήσετε ανοιχτέ διαδικασίε, δεν μπορείτε να, να κάνετε διάλογο, δεν μπορείτε να έχετε διαπραγματεύσει. Όχι, πολλά επιτρέπονται εντό αυτού του συστήματο. Ένα συγκεκριμένο παράδειγμα, πώ λειτουργεί αυτό στην πράξη. Έφερα μαζί μου ένα ε, μια σύμβαση εταιρική σχέση για έναν στην ε, στο Δήμο του Σίτιου, στην Νότια Δανία. Εδώ το Δημοτικό Συμβούλιο ακολούθησε τη διαδικασία των ε, δημοσίων συμβάσεων με διάλογο και διαπραγματεύσει. Η συμβάλλουσα αρχή από πολιτική άποψη ήταν πολύ ευαίσθητη σε αυτό το θέμα. Μιλάμε για ηλικιωμένου οι οποίοι θα έπρεπε να συμμετέχουν στη σύμβαση. Εδώ λοιπόν υπήρχε μια βασική διαδικασία, κάποιοι βασικοί όροι, αλλά ζητήθηκε από τους ιδιωτικούς ε, συμμετέχοντες να δώσουν ιδέες, ιδέες για το πώς θα μπορούσε να ανανεωθεί όλη αυτή η... όλο αυτό το εγχείρημα. Λοιπόν, εδώ υπήρξαν πραγματικά καινοτόμες λύσεις, η ίδια διαδικασία ήταν καινοτόμος και αυτό θα σας έλεγα να σκεφτείτε στη συνέχεια της διαδικασίας σας. Σας ευχαριστώ. Well, thank you very much indeed. Ευχαριστώ πολύ και εσάς και τους ε, προηγούμενους τρεις εμπειρογνώμονες. Ήταν πραγματικά ενδιαφέρον το υλικό που μας δώσατε. Είσαστε πράγματι εμπειρογνώμονες. Τώρα θα ήθελα όμως να ξεκινήσει η συζήτηση. Ο εισηγητής και οι σκιώδεις εισηγητές ε, να λάβουν το λόγο. Δεν ξέρω τώρα ο κύριος Σταραμπέλα, αν θέλει να λάβει το λόγο, οι ισχυώδεις συζητητές, απλώς θα ήθελα να δω αν θέλει κάποιος να θέσει ερωτήματα. Παρακαλώ να περιοριστείτε σε ένα λεπτό στις ερωτήσεις σας για να μπορέσω να, καλύψω, να καλύψουμε το χρόνο που χρειάζεται. Ο κύριος Κομφεράτη, η κυρία Βάιλερ, η κυρία Ρούλε, Σαλντεμόσε, ο κύριος Σβάμπ. Ένα λεπτό καθένα σας. Ενδεικτικά ένα λεπτό. Αν έχουμε δεύτερο χρόνο, μπορεί να, περισσότερο χρόνο μπορεί να επανέλθουμε. Κομφεράτη πρώτα. Ευχαριστώ. Άκουσα να γίνονται παραπομπές στο κόστος των διαγωνισμών. Προσπάθησα λοιπόν να σκεφτώ πώς θα λειτουργήσει αυτό με τη δεσμευτική λύση των κοινωνικών ε, κριτηρίων στα πλαίσια των δημοσίων διαγωνισμών. Συμφωνώ με την απέτηση να υπάρχει αυτού του είδους ε, η δέσμευση με κοινωνικέ προτεραιότητε. Όμω κάποια προσαρμογή θα πρέπει να γίνει, να είμαστε πολύ προσοχή, προσεκτικοί. Διότι μεταξύ διαφορετικών χωρών κάθε διαδικασία δημοσίων ε, προμηθειών έχει διαφορετική μορφή. Εάν γίνει ένα απόσπαστο μέρο ε, το κοινωνικό σκέλος των δημοσίων διαγωνισμών, δεν θα μπορούμε σε κάποιες περιπτώσεις να λειτουργούμε και με την αναζήτηση του χαμηλότερου κόστους. Βεβαίω η μείωση του κόστου οφείλεται και στην μερική ή τιμή εφαρμογή των κοινωνικών ρητών. Άρα το ένα μπορεί και να λειτουργεί ει βάρο του άλλου. Γι' αυτό πιστεύω, αλλά φαντάζομαι θα το σχολιάσουμε και μετά, ότι πρέπει στο βασικό σύνολο των κανόνων να έχουμε συγκεκριμένε διατάξει ό,τι αφορά την καταπολέμηση τη διαφθορά. Είναι, είναι τέτοια η κλίμακα των δημοσίων διαγωνισμών που προσελκύουν το οργανωμένο έγκλημα. Θα πρέπει λοιπόν τα μέτρα με τις κοινωνικές να μην τα θεωρούμε παράλληλα, διαφορετικά. Όχι, να είναι στο, στην καρδιά των ε, ρυθμίσεων που θα προβλέψουμε. Um, um, ο κύριος Έγγελ, γιατί είχε πει προηγουμένως ότι ήθελε να λάβει το λόγο. Ο οποίος είναι ο σκιώδης συγητής ε, για τη μεριά του ΕΛΚ. Αν θέλετε λοιπόν να θέσετε κάποια ερωτήματα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να σταθώ σε κάτι που δεν είναι κανονικά πάνω στην ημερήσια διάταξη, αλλά νομίζω ότι θα έπρεπε να παίζει κάποιο ρόλο. Χθε. Πήγα να οδηγήσω ένα αυτοκίνητο που ήταν αυτοκίνητο που λειτουργούσε με υδρογόνο. Δεν θα αναφέρω την ε, μάρκα του αυτοκινητού, γιατί αυτό δεν θα ήταν θεμητό. Απλώς, αυτό που θέλω να πω είναι αυτό το αυτοκίνητο είχε δανεικές πινακίδες. Ενώ χρησιμοποιείται στο Βελίο. Γιατί όμως. Η δυνατότητα για ένα τέτοιο αυτοκίνητο να έχει την τεχνική οργάνωση που χρειάζεται για να λειτουργήσει. Ε, η διαδικασία αυτή κράτησε 9 μέρες και μετά το αυτοκίνητο αυτό πήρε την έγκριση να κυκλοφορήσει. Στο Βέλιο θα χρησιμοποιήσει θα χρειαζόταν έξι μήνες. Με κάθε σεβασμό για τους Βέλγιους, με τους Βέλγους. Αν θεωρούμε ότι κάτι μπορεί να λειτουργήσει και να κυκλοφορήσει στους δρόμους της Δανίας, είναι τόσο επικίνδυνο να το εγκρίνουμε να κινηθεί στο Βέλγιο. Αυτό οδηγεί στο ερώτημα το οποίο θέλω να θέσω. Το θέμα της αμοιβαία αναγνώρισης μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για κάθε λογής πράγματα. Γιατί αν μιλάμε για κριτήρια περιβάλλοντος, αν μιλάμε για κοινωνικά κριτήρια, αν μιλάμε για ένα άλλο στοιχείο που συζητούσαμε τους εμπλεκομένους που είναι το δίκαιο εμπόριο και οι ετικέτες ε, δικαίου εμπορίου αναρωτιέμαι μήπως αντί να εφεύρουμε νέους κανόνες σε ευρωπαϊκό επίπεδο που είναι πολύ δύσκολο να, τους, ε, να συμμορφωθούμε με αυτούς και δύσκολο να τους καταλάβουμε και επειδή δεν υπάρχουν χρειάζονται πολύ προσπάθεια και σχεδιασμό μήπως θα ήταν απλούστερο να εξασφαλίσουμε ότι αν μας ενδιαφέρει πράγματι η εσωτερική αγορά και τα 60 χρόνια ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης που έχουν περάσει, θα πρέπει να μας σε θέση να πούμε σε όλους αυτούς τους τομείς αν ένα προϊόν, μια υπηρεσία, ένας πάροχος υπηρεσιών, ένας παραγωγός σέβεται κριτήρια που ισχύουν σε ένα κράτος μέλος, τότε οποιαδήποτε κριτήρια τα οποία θεσπίζονται σε ένα άλλο κράτος μέλος θεωρούνται ότι καλύπτονται μέσα από την έγκριση σε μια άλλη χώρα. Δεν το έχουμε συζητήσει αυτό, αλλά δεν ξέρω αν αυτό θα έκανε τη ζωή μας ευκολότερη. Ως εισηγητής για την έγκριση κυκλοφορείς αυτοκινήτων, θα, πω κάτι, θα σου πω κάτι ιδιωτικά μετά, αλλά αύριο συζητάμε και τα πρότυπα που είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Κυρία Βάιλαρ έχει το λόγο μετά. Κύριε Πρόεδρε, ξανάρχομαι στο δίκαιο συμβάσεων και το δίκαιο απονομής συμβάσεων. Έχω ένα ερώτημα προς την κυρία Βερόνη Καλίσεν και ένα ερώτημα προς τον κύριο Σάρφ, τον Ιάκοπ Σάρφ. Κύριε Σάρφ, Νομίζω ότι σε σχέση με τα κοινωνικά κριτήρια κάπως φάσκεται και αντιφάσκεται. Αυτό που είπατε το τελευταίο παράδειγμα είναι πολύ σωστό και είναι πολιτικά ε, επιθυμητό επίσης. Αλλά είπατε όλα αυτά όπου, όπου έχει νόημα. Και αυτό το υποστηρίζω. Όπου πράγματι έχει νόημα. Νομίζω ότι είναι καιρό να εισαγάγουμε, να περισσότερα τα κοινωνικά κριτήρια από ό,τι στο παρελθόν. Και γι' αυτό έρχομαι στο ερώτημα που θέλω να θέσω στη Βερόνικα Νίλσεν. Στην Γερμανία έχουμε κάποια κρατήδια τα οποία έχουν νομοθεσία για την ε, απονομή συμβάσεων όπου περιλαμβάνεται το ότι πρέπει να υπάρξει σεβασμός των ε, συλλογικών συμβάσεων αλλά υπάρχουν σε άλλη νομοθεσία ότι μία σύμβαση θα πρέπει να έχει το πολύ 20% εργαζόμενους κατά πόσπαση. Σε όλους αυτούς τους τομείς θα μπορούσε αυτό να ισχύει μονάχα για τη Γερμανία μια τέτοια λογική και όχι για άλλα κράτη-μέλη. Θεωρείτε ότι θα είχε νόημα να εισαγάγουμε τέτοιες ρυθμίσεις και σε ευρωπαϊκό επίπεδο χωρίς να έχουμε προηγουμένως ένα συνεκτικό πλαίσιο για την ε, κατακύρωση συμβάσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ευχαριστώ η κυρία Ρούλα. Και εγώ συμφωνώ με τους συζητητές ότι το θέμα του πώς αγοράζουμε κάτι και όχι τι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Για, το, για τα άλλα πρέπει να βρούμε διαφορετικά εργαλεία. Εμάς μας ενδιαφέρει η νομοθεσία στα θέματα αυτά. Έχουμε ακούσει από πολλά κράτη-μέλη ότι υπάρχουν προβλήματα για τα θέματα αυτά. Επίση υπάρχει το θέμα τη καινοτομία που θέλουμε να προωθήσουμε. Γνωρίζουμε τι γίνεται σε άλλε περιπτώσει. Παραδείγματο χάρη οι Δήμοι τη Σουηδία που δεν μπορούν να αγοράσουν, παραδείγματο χάρη, κρέα από ζώα τα οποία κρατούνται, εκτρέφονται σε ορισμένε συνθήκε και του απαγορεύεται αυτό από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Νομίζω ότι εδώ η Τζάνετ Ρίτσαρτ έχει δίκαιο ότι μπορούμε να γίνουμε υπερβολικοί στην λεπτομεριακή ρύθμιση και ουσιαστικά να διαθρέψουμε, να εκθρέψουμε μια γραφειοκρατία και όχι να πετύχουμε αυτό το οποίο θέλουμε. Δηλαδή να αφαιρέσουμε από τις αρχές οι οποίες παίρνουν την απόφαση να χρησιμοποιήσουν και την κρίση τους. Γι' αυτό θέτω ένα ερώτημα σε εσά. Όπως είπατε, είναι σημαντικό να υπάρξει κάποια επιρροή στα θέματα της νομοθεσίας, αλλά θα ήθελα να σταθώ στο θέμα της στοχοθεσίας και της απλοποίησης. Πώς μπορείτε να εξασφαλίσετε μια ε, ισορροπία μεταξύ των δύο αυτών, γιατί αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Ευχαριστώ. Η κυρία Σόλντε Μόζε έχει το λόγο. Και εγώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ένα ερώτημα έχω για τον κύριο Σάφ. Νομίζω ότι είδα στην παρουσίασή του, άκουσα κάτι για τα όρια, για τα κατόφλια αλλά δεν τα ανέφερε. Τι εννοείται με αυτό. Πρέπει να είναι πιο ψηλά, πιο χαμηλά ή αυτά που υπάρχουν. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Σβάμπ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μετά από αυτό που είπε ο κύριος Κομφεράτη, θα ήθελα να δώσω συνέχεια στο σημείο αυτό. Όταν μια προκήρυξη περιλαμβάνει ορισμένα κριτήρια πρέπει όλοι οι υποβάλλουν προτάσεις να εκπληρούν αυτά τα κριτήρια. Αλλιώς αποκλείονται από το διαγωνισμό. Επομένως, τα κριτήρια τα οποία προβλέπονται κάθε φορά θα πρέπει να τηρηθούν από όλους τους ανταγωνιζόμενους. Το σημαντικό ερώτημα όμως είναι, όπως είπε και η κυρία Ρούλε, πώς θα εξασφαλίσουμε ότι τα κριτήρια τα οποία είναι δυνατόν να τεθούν θα καθοριστούν με τρόπο σαφή και ασφαλή ώστε έχουν σαν αποτέλεσμα να εξασφαλίσουν μια αποτελεσματική διαφοροποίηση της διαδικασίας παραγωγής. Δηλαδή να πετύχουν το στόχο αυτό που θέλουμε στην παραγωγή μέσα από τις τεχνικές λοιπόν αυτές ε, προδιαγραφές να κατευθύνουμε προς μια κατεύθυνση την παραγωγή. Νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να έχει μια προτεραιότητα εναντί άλλων εξωτερικών κριτηρίων στη διαδικασία επιλογής, αλλά από την άλλη πλευρά και εδώ αναφέρομαι σε αυτό που είπε ο κύριος Κομφεράτη, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται σαν πρόσχημα για να αποκλείονται τεχνιέντος ορισμένοι που διαγωνίζονται. Ευχαριστώ. Αν κάποιος άλλος δεν θέλει να λάβει το λόγο, <clears throat> κυρία Γκέπχατ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ θέλω να θέσω ένα ερώτημα στην κυρία Νίλσεν, γιατί αναφερθήκατε στα κοινωνικά κριτήρια, τα οποία για μας έχουν μια πολύ μεγάλη σημασία. Έχω τονίσει στο παρελθόν ότι χρειαζόμαστε μεγαλύτερη σαφήνεια δικαίου, γιατί πολλέ φορέ υπάρχει μια ασάφεια για το ποια είναι τα κοινωνικά κριτήρια τα οποία πρέπει να εφαρμοστούν και τι ανήκει στο. Μάλκο Μποζακρί στο μικρόφωνο σου. Να έχουμε λοιπόν μεγαλύτερη σαφήνεια και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και ε, πρέπει. Αλλά έχω και την εντύπωση και εδώ έρχομαι στο ερώτημά μου Όταν προσπαθούμε να κάνουμε σαφέστερα τα κριτήρια και δεν ξέρω ότι μπορούμε να το πετύχουμε αυτό πάντα, αυτό σημαίνει ότι περιορίζουμε τη δυνατότητα εφαρμογής των κοινωνικών κριτηρίων σε σχέση με το παρελθόν. Και αυτό δεν μου φαίνεται σωστό. Εγώ πιστεύω αντίθετα ότι θα πρέπει να επιζητήσουμε να εξασφαλίσουμε ότι οι αποφάσεις και το ευρωπαϊκό δίκαιο για τα κοινωνικά θέματα να ενισχυθεί με αυτών των διαδικασιών και όχι να αποδυναμωθεί. Αυτό θα ήταν αποφασιστική σημασία για μένα και επίσης θα ήθελα να επανέλθω στο θέμα των εργολαβιών και υπ εργολαβιών. Είναι απόλυτα σημαντικό να λαμβάνονται αυτά τα κριτήρια και στις υπεργολαβίες και επομένως να υπάρχει μια δεσμευτικότητα των κριτηρίων αυτών για τους υπεργολάβους και τους υπυπεργολάβους. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Μάλκομ. Έχω άλλους δύο μιλητές, αν σύντομοι, η κυρία Βανιού, η κυρία Φερχέιν. Θα είμαι σύντομη, γιατί η κυρία Γκέμπαρτ νομίζω ότι ανέφερε τουλάχιστον το μεγαλύτερο μέρος της ερωτήσεώς μου. Θέλω να θέσω το ερώτημα στην κυρία Νίλσεν πώς θεωρείτε ότι είναι δυνατόν να σέβεται κανείς τις συλλογικές συμβάσεις κάθε κράτους και συγχρόνως να αποφέρει τους κινδύνους κοινωνικού ντάμπινγκ αν δεν υπάρχει μια ε, αλυσίδα ευθύνης για τους, εργολάβους, για τους υπεργολάβους των δημοσίων προμηθειών. Κύριε Βερχάιεν. Και εγώ θέλω να θέσω ένα ιδιαίτερο ερώτημα προς τον κύριο Ιάκοπ Σαφ. Αναφερθήκατε για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τις δυσκολίες που έχουν να αντιμετωπίσουν λόγω της πολυπλοκότητας του δικαίου προμηθειών. Αντίστοιχο είναι το πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουν και οι μικρομεσαίοι δήμοι, οι οποίοι πολλές φορές έχουν να αντιμετωπίσουν πολύ μεγάλη πολυπλοκότητα και δεν μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτές τις διαδικασίες και προκύπτουν με τον τρόπο αυτό πάρα πολλά σφάλματα. Βλέπετε λοιπόν ότι η αναθεώρηση οδηγεί σε κάποια βελτίωση ή παραμένουν τα πράγματα εξίσου ε, πολύπλοκα. Θέλετε να δημιουργηθεί περισσότερη ευελιξία στα θέματα αυτά. Πώς βλέπετε να αξιολογούν οι επιχειρήσεις την πρόταση της Κομισιόν. Επίσης μιλήσατε για ιδιαίτερες κοινωνικού χαρακτήρα εταιρικέ σχέσεις μεταξύ Δήμων και κοινοτήτων από τη μια μεριά και επιχειρήσεων. Και αυτό πάλι θα οδηγήσει σε δυσκολίες όταν κάνει κάτι τέτοιο σε ό,τι αφορά την ισότητα ευκαιριών στους δημόσιους διαγωνισμούς. Πολλές φορές οι μικρομεσαίοι δήμοι αποτρέπονται να επιλέξουν επιχειρήσεις που τηρούν τα κοινωνικά κριτήρια ή δίνουν την καλύτερη αξία σε σχέση με το κόστος γιατί φοβούνται ότι θα προκύψει κάποια νομική προσφυγή εναντίον τους και επομένως προσπαθούν να αποτρέψουν κάτι τέτοιο. Είναι και αυτό ένα τμήμα του προβλήματος για σας ή όχι. Σας ευχαριστώ για αυτά τα ερωτήματα πολύ χρήσιμα. Τώρα θα δώσουμε το λόγο στους εμπειρογνώμονές μας για να απαντήσουν ιδιαίτερα τον κύριο Σαφ αλλά και την κυρία Νίλσον Δύο λεπτά τον καθένα για να απαντήσετε. Αν έχετε πολλές απαντήσεις βέβαια θα το σεβαστούμε, αλλά προσπαθήστε να σεβαστείτε το δίλεπτον. Ο κύριος Σάρφ πρώτος. Ευχαριστώ. Τα όρια και τι φρονώ για αυτά. Εμείς θεωρούμε ότι τα ισχύοντα όρια είναι πολύ χαμηλά. Και για τις επιχειρήσεις αυτό σημαίνει υψηλότερο διοικητικό κόστος. Εδώ μιλάμε για προσφορές όπου που ποτέ δεν είναι διαμεθοριακές οι προσφορές. Προτείνουμε λοιπόν πολύ ψηλότερα όρια γιατί από επιχειρησιακή απόψεως αυτό θα μείωνε το κόστος των διαγωνισμών. Δεν θέλουμε να υπάρξει μία μαύρη τρύπα όπου, βέβαια, όπου θα πέφτουν αυτόματα όλα τα συμβόλαια. Απλώς μία απλοποίηση, ένα ελαφρύτερο καθεστώς. για τη γενικότερη αξιολόγηση της οδηγίας από επιχειρησιακής πάντοτε απόψεως νομίζουμε ότι μπορεί να βελτιωθεί πολύ από απελευθέρωση. Εκατό σελίδες είναι πάρα πολλές. Ο ισχύων δανεικός νόμος για τις προμήθειες είναι μία σελίδα, μία. Και υπάρχει βέβαια πολλή νομολογία από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Αλλά συγκρίνουμε μία σελίδα με 100. Δεν χρειαζόμαστε αναγκαστικά περισσότερους κανόνες. Ιδιαίτερα δε για την πράσινη προσφορά. Η Δανία, η Σουηδία κτλ. ήδη απλοποιούν τους κανόνες για τα κοινωνικά καριτήρια, εγώ σας είπα να χρησιμοποιηθούν μεν οι κοινωνικοί εταίροι αλλά όχι συγκεκριμένα και απαραίτητος για τις προμήθειες. Δεν χρειάζεται δηλαδή να συσχετιστεί γενικά η συνεργασία και με τις προμήθειες. Δεν πιστεύω λοιπόν ότι θα διευκολύνει τα πράγματα να υπάρξει μια ενωσιακή διευθέτηση με περισσότερα κοινωνικά κριτήρια. Δεν νομίζω καν ότι γίνεται αυτό γιατί και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και η τοπική αυτοδιοίκηση δολοφονούνται από τέτοιου είδους κεντρικές διευθετήσεις. Ευχαριστώ. Η κυρία Νίλεσον. Ευχαριστώ. Οι ερωτήσεις προς εμένα έμοιαζαν πολύ. Ήταν όλες για τα κοινωνικά κριτήρια. Πρέπει να διαχωρίσουμε εδώ από τη μια τα κοινωνικά κριτήρια που είναι απολύτως δεσμευτικά και τα άλλα που είναι προαιρετικά. Βασικά οι συνθήκες εργασίας, οι συλλογικές συμβάσεις κλπ. πρέπει να είναι υποχρεωτικές και να γίνονται σεβαστές. Προβλέπεται να γίνονται σεβαστές αλλά δεν είναι πάντοτε. Και να είναι υποχρεωτικό αυτό για όλη την αλυσίδα Άλλα κριτήρια όμως, που και αυτά αναφέρθηκαν όπως η δημιουργία ειδικών θέσεων για μακροχρόνιους ανέργους κλπ. Αυτά μπορούν να μην είναι τόσο υποχρεωτικά αλλά πυροαιρετικά. Για μένα λοιπόν υπάρχει μια διαφορά το θέμα είναι μέχρι ποιου σημείου είμαστε διατεθειμένοι να πάμε για τα κοινωνικά, με τα κοινωνικά κριτήρια, εθνικά πρότυπα, τα κτλ. Κάτι που ακούστηκε και το βρίσκω σωστό είναι ότι πρέπει να προσέξουμε το εύρος εφαρμογής της οδηγίας να μην είναι πολύ περιορισμένο όταν ορίζονται τα κριτήρια. Όσο για το συγκεκριμένο, για τους μερικώς και προσωρινώς εργαζομένους, δεν ξέρω αν υπάρχουν τέτοια κριτήρια και για αυτούς σε μερικές χώρες ή όχι. Θα το ελέγξω. Ίσως η Γερμανία εφαρμόζει και να τα πει ο Γερμανός συναδέλφος γιατί εγώ δεν τα ξέρω. Θα το ελέγξω πάντως. Αν δεν απατώμε, αυτά είχα να πω. Πρίτσαρντ. Ευχαριστώ. Ήθελα να απαντήσω στην ερώτηση της κυρίας Ρούλε για το πώς θα μπορούσε να πλουστευτεί περαιτέρω η οδηγία. Πολλά παραδείγματα θα μπορούσα να δώσω. Ένα, λόγου χάρη, για το πώς οι οδηγίες έχουν κοιτάξει τις επιλογές των κριτηρίων και εάν θα πρέπει η απόφαση να λαμβάνεται βάσει της τιμής, της χαμηλότερης τιμής, του κόστους, την ελκυστικότερη από οικονομικής άποψης ε, προσφορά, την ε, αντιστοιχεία κόστους, τιμής δηλαδή και αξίας. Εδώ λέμε σήμερα ότι πρέπει να φύγουμε από το κριτήριο της χαμηλής τιμής μόνον και να κοιτάξουμε κατά πόσον μπορούμε να εμπλουτίσουμε την άποψη ότι χρειαζόμαστε περισσότερη αξία για την ίδια τιμή. Το χαμηλότερο κόστος είναι ένα κριτήριο, αλλά νομίζω εδώ η επιθυμία ήταν να ενθαρρυνθεί το κόστος του κύκλου ζωής στα πλαίσια της ανάθεσης ε, συμβάσεων και της σχετικής απόφασης μεταξύ των προφορών, προσφορών. Όμως, ο τρόπος που έχει καταρτιστεί η πρόταση προκαλεί σύγχυση. Δεν επιτρέπει απλώς η διαδικασία δημόσιων προμηθειών να αξιοποιήσει σωστά το εργαλείο και να το αναπτύξει περαιτέρω και να το προσαρμόσει όπως χρειάζεται, αλλά προκαλεί σύγχυση. Δηλαδή, μόνο όσα μπορούν σε νομισματικού όρου να τεθούν ε, επιτρέπουν τη χρήση αυτού του κριτηρίου. Όπω σωστά είπε και ο κύριο ε, Αλμπάνο, το κόστος, ε, εφόσον αποσβεθεί σε ένα χρονικό διάστημα, δίνει τελικά μεγαλύτερο όφελος στον αγοραστή, αλλά δεν είναι σαφές ότι οι υπεργολαβίες έχουν λαθεί ληφθεί υπόψη. Θα έπρεπε όμως να μπορούν να συμπεριλαμβάνονται. Διότι είναι ένα στοιχείο για καλύτερη αξία και αυτό θα είναι ένας απλούστερος τρόπος να το εκφράσουμε. Για να περάσουμε από τη χαμηλότερη αξία στην ε, καλύτερη, χαμηλότερη τιμή μάλλον, στην καλύτερη αξία. Ίσως χρειάζεται προσεκτικότερη διατύπωση. Πάλι ξεπέρασα το χρόνο μου. Εάν μπορείτε πολύ γρήγορα να μας συμπληρώσετε. Ναι, για τα κοινωνικά κριτήρια. Και το κατά πόσον πρέπει να επιδιώξουμε ποιότητα στα κοινωνικά κριτήρια το πεδίο. Το πεδίο αυτό να είναι πιο συγκεκριμένο. Κάποιες παρατηρήσεις που έκανε ο κύριος Σάρφ βλέπουμε ότι όπου οι καλύτερες πρακτικές προχώρησαν, φιλόδοξοι, οι πιο ικανοί από όσους λειτουργούν στην πράξη, κατάφεραν να κάνουν αυτό που ήθελαν χωρίς περιορισμούς. Υπάρχουν πολλέ προκλήσει. Το πώ να αντιμετωπίσουμε τα κοινωνικά κριτήρια με διαφανή τρόπο. Όμω θα πρέπει η αρχή τη διαφάνεια να είναι σαφή εξ αρχή και μετά να αναπτυσσούμε όλο και περισσότερο τα υπάρχοντα η, ισχύουσα και η προτινόμενη οδηγία είναι πολύ αυστηρές για την ε, δυνατότητα συμπερίληψης κοινωνικών κριτηρίων. Ευχαριστούμε ο Δ. Αλμπάνο τελευταίος. Ευχαριστώ να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία να βρίσκομαι εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο και αν ε, μου επιτρέπετε να μιλήσω τελικά για να απαντήσω σε μια από τις βασικές ανησυχίες. Κύριε Κοφεράτη, Εσεί εκφράσατε μια μεριμνά για τις δημόσιες προμήθειες. Νομίζω το πλέον σημαντικό που θα πρέπει να έχουμε υπόψη είναι ότι τη στιγμή που αναδίθεται μια δημόσια σύμβαση. Πολλές φορές αξίζει και εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ η σύμβαση αυτή, αλλά βάσει υποσχέσεων. Άρα οι αναθέτουσες αρχές το επόμενο δευτερόλεπτο μετά την επιλογή και την ε, ανάθεση ξεκινάει η δουλειά τους. Θα μπορούσαν να υπάρχουν κάποιε ελάχιστε απαιτήσει λοιπόν περιβαλλοντικά, κοινωνικά κριτήρια, αλλά το πραγματικό πρόβλημα είναι το πρόβλημα της επαληθευσιμότητας των υποσχέσεων και όσων έρχονται να ακολουθήσουν από την επιχείρηση που ανέλαβε τελικά τη σύμβαση. Αυτό νομίζω που έθιξε ο κ. Κοφεράτη ήταν ιδιαίτερα σημαντικό, διότι ακριβώ αυτή τη στιγμή, εάν έχει κανείς συνείδηση ότι υπάρχει παράγοντα κινδύνου το επόμενο ακριβώ δευτερόλεπτο που μπορεί να κρατήσει και για χρόνια κατά την εκτέλεση τη σύμβαση, αυτό δημιουργεί όλε όλες τις πιθανότητες ε, της διαφθοράς λόγω χάρη που δεν ε, καταπολεμάται αν προσθέσουμε αυστηρότερες διατάξεις ή κανόνες. Ίσα ίσα μπορούμε να αποκρούσουμε την διαφθορά όχι με πρότυπα που θα επικαλύπτονται και πολλές φορές αντιφάσκουν, αλλά όπως έλεγε και η Συνάδελφο, με την οποία συμφωνώ απολύτως, με καλύτερες πρακτικές, με τα παραδείγματα που έχουν λειτουργήσει στην πράξη, με την ανάθεση ευθυνών, με απόδοση κινήτρων, με την ε, δημόσιο διδολογικό κώδικα που δεν υπάρχει σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Μόνον κατά αυτόν τον τρόπο θα ανακτήσουμε την συνέπεια μεταξύ του τι γίνεται πριν και τι μετά, το εξάντε και το εξπόστ. Έτσι, τα κοινωνικά, τα περιβαλλοντικά κριτήρια κατά κάποιο τρόπο γίνονται πολιτική επιλογή και αυτό είναι και η ουσία τους. Όμως το σημαντικό είναι να μεταφραστεί ο πολιτικός στόχος σε πρακτική εφαρμογή. Και αυτό θα μπορούσε να παραμείνει κενό γράμμα. Ευχαριστώ. Well, thank you. Ευχαριστώ πολύ λοιπόν και τους τέσσερις ε, ε ομιλητές. Θα ήθελα τώρα να περάσουμε στη δεύτερη φάση της ε, μας και προηγουμένως θα ήθελα να καλωσορίσω τον Κλάους Βίτνερ, ο οποίος είναι ο Διευθυντής ε, της Μονάδος για την Εσωτερική Αγορά. Χαίρομαι που είσαστε εδώ και ελπίζω ότι αν έχουμε εξοικονόμηση χρόνου θα σας δώσουμε τη δυνατότητα να πείτε δύο λόγια στο τέλος και έχουμε επίσης δύο από τους συντάκτες γνωμοδότησής μας εδώ γιατί θα έχουμε γνωμοδοτήσεις ο κ. Σούστερ από την Επιτροπή Εξωτερικού Εμπορίου και ο κ. Μπαλτσάιτζης από την Επιτροπή Βιομηχανίας. Ερχόμαστε λοιπόν. Υπάρχουν άλλοι και ο κ. Στοσάια από την Επιτροπή Απασχόλησης, βεβαίως. Προχωρούμε τώρα στα επόμενα θέματα, στο επόμενο θέμα. Συζητήσαμε για τα θέματα της απλοποίησης και της ε, εποπτείας εφαρμογής. Ερχόμαστε λοιπόν στο θέμα αυτό τη απλοποίηση, Δίνω το λόγο στην κυρία Αγγέλη Καπόθ Μούργελε, που είναι διευθυντή σε θέματα πολιτική στο Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Δήμων και Περιφερειών και η οποία έχει μια ιδιαίτερη εμπειρία για τα θέματα αυτά και εκπροσωπεί πολλέ ε, αναθέτουσες αρχέ ε, ευρωπαϊκών δήμων και περιφερειών και μπορεί να μα πει κάτι περισσότερο για τα θέματα αυτά τη απλοποίηση. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε αγαπητά μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κυρίε και κύριοι. Πρέπει να σας πω ότι δεν είχαμε την ευκαιρία να διαβουλευτούμε πριν από τη συνάντηση αυτή, αλλά αυτά που είπε ο Δανός συνάδελφός μου αντανακλά πάρα πολύ την εμπειρία των τοπικών και περιφερειακών αρχών που εκπροσωπεί το δικό μας συμβούλιο, το ΣΕΜΡΑ. Είμαστε μια ευρωπαϊκή οργάνωση που καλύπτει όλες αυτές τις ε, οργανώσεις δήμων και κοινοτήτων και έχουμε υπό την αιγύδα μας 60 τέτοιες οργανώσεις. Χαιρόμαστε πάρα πολύ για την ευκαιρία που έχουμε να λάβουμε το λόγο σήμερα σαν εκπρόσωποι των τοπικών και περιφερειακών αρχών, γιατί οι οδηγίες αυτές για τις δημόσιες συμβάσεις είναι πολύ σημαντικές για τα μέλη μας και όπως ξέρετε ένα πολύ μεγάλο μέρος των δημοσίων συμβάσεων γίνεται σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο και όχι μόνο σε εθνικό τα τελευταία χρόνια η εμπειρία μας είναι ότι γίνονται όλο και πιο πολύπλοκες οι διαδικασίες σύναψη συμβάσεων, δύσκολες στην εφαρμογή τους, πολυδάπανες και δύσκολες στην εφαρμογή τους. Και για τους, αυτούς που υποβάλλουν προσφορές και για τις αρχές που απονέμουν τις συμβάσεις. Γι' αυτό το CMR έχει δημοσιεύσει ένα έγγραφο για την ε, χρήση ε, των δημοσίων συμβάσεων ε, και τα προβλήματα που παρουσιάζουν. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια μετακίνηση από τον στόχο της αξίας σε σχέση με το κόστος σε συμβόλαια τα οποία μπορεί να είναι πιο πολυδάπανα αλλά εξασφαλίζουν νομική ασφάλεια. Ξέρουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση συμμερίζεται πολλά από, τα, από τις ανησυχίες μας. Το, το ψήφισμα του 2011 του Κοινοβουλίου τόνισε την ανάγκη απροποίηση των κανόνων συγκεκριμένα. Εγώ θέλω να αντιμετωπίσω δύο θέματα σήμερα. Το ένα είναι η απλοποίηση και το άλλο είναι η συνεργασία σε δημόσιο επίπεδο σε σχέση με, τους, με τις συμβάσεις αυτές. Η πρόταση της Κομισιόν από το Δεκέμβριο του 2011, κατά την άποψή μας, δεν επιτυγχάνει το στόχο της απλοποίησης, κάθε άλλο. Ξεπερνάει τα όρια αυτού που μπορούμε να θεωρήσουμε αναλογικό και σε μεγάλο βαθμό αντιβαίνει και προς την αρχή της επικουρικότητας το σχέδιο οδηγία έχει πάρα πολύ λεπτομεριακέ ρήτρε για, μια σειρά θεμάτων που κατά την άποψή μα δεν πρέπει να τύχουν ρύθμιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο σε τέτοιο βαθμό. Υπάρχει μια κόποση που προέρχεται από υπερβολικά λεπτομεριακέ ρυθμίσει σε ευρωπαϊκό επίπεδο και αυτό το οποίο χρειαζόμαστε είναι λιγότερη και όχι περισσότερη διαχείριση και ρύθμιση. Αυτό το έδειξε και το τελευταίο Συμβούλιο το Ιαρινό Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 1 και 2 Μαρτίου του 2011 που τόνισε, συγγνώμη, που τόνισε ότι πρέπει να συνεχιστεί η προσπάθεια μείωση του διοικητικού και ρυθμιστικού άγχου σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Θέλουμε να έχουμε στόχου κατά τομής και πιστεύουμε ότι η πρόταση για τι δημόσιε συμβάσει θα ήταν μια ευκαιρία για τον Ευρωπαίο νομοθέτη να θέσει ένα χρήσιμο παράδειγμα. Να σα δώσω μερικά παραδείγματα νέου άχθους που προβλέπεται από αυτό το κείμενο. Ε, υποχρεώσεις δημοσιοποίησης για κοινωνικές και άλλες υπηρεσίες. Νέε διαδικασίε σε εθνικό επίπεδο για αυτέ τι υπηρεσίε άρθρο 76. Δημιουργία νέων εποπτικών φορέων σε εθνικό επίπεδο, άρθρο 84. Πρόσθετες εξηγήσει σε σχέση με την αξία του συμβολέου, που, του, της συμβάσεως που επιλέγεται, άρθρο 44. Επαχθείς ανάγκε για εκθέσει και κοινοποιήσει προ την Κομισιόν, Αρθρο 32, 85 και 86 και τέλο νέες διαδικασίες συμβάσεων σε σχέση με δανειακές υπηρεσίες, άρθρο 10, δέλτα, και νέες διαδικασίες για τις νομικές υπηρεσίες. Όλα αυτά πιστεύουμε ότι είναι υπερβολικά και στρέφονται κατά της αρχής της επικουρικότητας. Χρειαζόμαστε, όπως είπε και ο Δανός ε, ομολογός μου, λιγότερες από 246 σελίδες ρυθμίσεων, όπως προτείνεται, όχι περισσότερες. Θεωρούμε λοιπόν επίσης ότι η οδηγία δεν είναι αποτέλεσμα εφιάς ρύθμισης που ήταν ένας στόχος της Κομισιόν στο παρελθόν. Επίσης κάποιες από τις ρυθμίσεις έχουν το χαρακτήρα εφαρμοστικών κατευθυντήριων γραμμών και δεν πρέπει να είναι τμήμα ενός νομοθετικού κειμένου. Τέτοια στοιχεία θα μπορούσαν να βρίσκονται σε ένα εγκόλπιο ή εγχειρίδιο που επιτρέπει ταχείες τροποποιήσεις εν καιρό για να παρακολουθήσει την εξέλιξη του τη νομοθεσία για τη σύμβασή Ζητούμε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λοιπόν και τα κράτη-μέλη να έχουν μια ευρεία προσέγγιση και να ακυρώσουν, να διαγράψουν όλε τι ρήτρε που είναι ιδιαίτερα λεπτομεριακέ. Οι τοπικέ και οι περιφερειακέ αρχέ υποστηρίζουν ιδιαίτερα την ανάγκη να υπάρχει ανοιχτό ανταγωνισμό και την ανάγκη να δημιουργεί ένα σαφέστερο καθεστώ, ένα πλέον καθεστώ, μάλλον ιδιαίτερα για τι μικρόμεσέ επιχειρήσει. Οι δημόσιε αρχέ υποστηρίζουν την αρχή τη συνθήκη για ισότητα, διαφάνεια και μη διάκριση αλλά το να εφαρμοστούν με τρόπο συνεκτικό οι πολύπλοκοι κανόνε των ευρωπαϊκών οδηγιών και των ευρωπαϊκών χρονοδιαγραμμάτων, χωρί να υπάρξει καμία προσφορά από παρόχου ε, προϊόντων και υπηρεσιών σε άλλα κράτη-μέλη, σημαίνει ότι είναι σπατάλη πόρων και χρόνου. Το πολύπλοκο αυτό καθεστώ δεν είναι αναλογικό με τα αποτελέσματα τα οποία επιτυγχάνονται. Πώς να έχουμε απλοποίηση στα θέματα αυτά. Υπάρχουν διαφορετικέ προσεγγίσεις. Πρώτα απ' όλα, όπως είπε ο προλαλής σας, μπορούμε να αυξήσουμε τα κατόφλια για αγαθά και υπηρεσίες. Αυτό θα βοηθούσε πάρα πολύ να μειώσει το χρόνο και το κόστος που δαπανάτε και από την πλευρά αυτών που υποβάλλουν προσφορές και από αυτή την πλευρά των αρχών απονομής. Δεύτερον, θα μπορούσαμε να έχουμε μια οδηγία πλαίσιο που να βασίζεται στις αρχές της ε, συνθήκης. Έχουμε την Συμφωνία Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, που με τα 24 άρθρα του δίνει ένα τέτοιο πολύ ελαφρό καθεστώς και είναι πολύ πιο ευέλικτο. Και επειδή πρέπει να υπάρχει συνεκτικότητα του πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΠΟΕ, θα πρέπει να ενθαρρύνουμε τον νομοθέτη να προσαρμόσει τις ευρωπαϊκές ρυθμίσεις αυτές του ΠΟΕ. Τρίτον, πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη συνειδητοποίηση και μεγαλύτερα κίνητρα για να βλέπουμε, για να προσπαθούμε να έχουμε καινοτόμε λύσεις, ιδίω στην ηλεκτρονική διαδικασία συμβάσεων. Ζητούμε λοιπόν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να πάρει μια τολμηρή στάση και να υποστηρίξει τις καινοτόμες αυτές λύσεις με ένα ελαφρό καθεστώς για τις ε, ευρωπαϊκές συμβάσεις. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε καταφέρει με τις κυρώσεις να περιορίσουμε και να επιτύχουμε το στόχο που θέλαμε, ας χρησιμοποιήσουμε μια οδό η οποία βασίζεται στην παροχή κινήτρων, θετικών κινήτρων για τις δημόσιες αρχές. Για μας είναι απαραίτητο οι δημόσιες αρχές να συνεργαστούν για να μπορέσουν να έχουν δημόσιε δημόσιες υπηρεσίες. Διακοινωτικές ή άλλες ε, υπηρεσίες δεν υπόκεινται στην οδηγία αυτή για τις ε, συμβάσεις και πρόσφατα το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο <clears throat> έδωσε μια διευκρίνηση για το θέμα αυτό που ήταν πάρα πολύ σαφή. Επιπλέον το άρθρο 11,4 δίνει την ερμηνεία της ε, Κομισιόν για την ομολογία του, του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, αλλά αυτό δεν πρέπει να αποτελέσει τμήμα τη οδηγία. Πιστεύουμε ότι η πρόταση αυτή περιλαμβάνει μια πάρα πολύ περιστατική ερμηνεία τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Θεωρεί ότι τα αμοιβαία δικαιώματα και υποχρεώσει είναι μια αποφασιστική προπόθεση η οποία πρέπει να χρησιμοποιηθεί για να αποκλείεται η συνεργασία δημόσιου τομέα με δημόσιο τομέα. Αλλά με τον τρόπο αυτό αφήνει πολλέ πλευρέ αυτή τη συνεργασία ανοιχτή. Είναι πάρα πολύ περιοριστική αυτή η διαδικασία των αμοιβαίων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων. Δεν καλύπτει τι τωρινέ πρακτικέ και μπορεί να τύχει κατάχρηση. Και αυτό, αυτές οι αναγκαιότητες δεν εμφανίζονται στην περίφημη υπόθεση στα Dranningu Hamburg 4806 και επομένως δεν θα έπρεπε να κωδικοποιηθούν με τον τρόπο αυτό. Δεν έχει νόημα λοιπόν να ε, γίνεται επίσης κάτι τέτοιο όταν, δεν, όταν δημιουργείται μια νέα νομική οντότητα για να αντιμετωπίσει το θέμα αυτό. Επομένως δεν μπορεί να υποχρεωθεί κανείς να έχει αυτή την αμοιβαιότητα. Πρέπει να υπάρξει μια προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η οποία να βασίζεται στην ισότητα και να ευθυγραμμίζεται με την απόφαση του δικαστηρίου στην περίπτωση στα Χάμπουργκ. Πιστεύουμε λοιπόν ότι πρέπει η διατύπωση να αντανακλά την ομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και να χρησιμοποιηθεί μέσα στο κείμενο της οδηγίας. Αυτή η οδηγία θα πρέπει να τονίζει ότι το θέμα αυτό της ε, μεταφοράς καθηκόντων μεταξύ δημοσίων οργανισμών είναι θέμα της εσωτερικής δίκης των κρατών μελών και όχι αντικείμενο των κανόνων συμβάσεων. Ελπίζουμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα παραμείνει πιστό στο ψήφισμά του του Οκτωβρίου 2011 Εν κατακλείδη, θέλω να σας περάσω τις προσδοκίες των τοπικών και περιφερειακών αρχών ότι θα πρέπει αυτές οι νέες ρυθμίσεις να κάνουν ευκολότερες τις δημόσιες συμβάσεις και όχι πιο πολυδάπανες και πιο πολύπλοκες και για αυτούς που υποβάλλουν προτάσεις και τις αρχές απονομές. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πραγματικά για την σαφέστατη αυτή παρουσίαση και για τις υψηλές αυτές προσδοκίες ε, προς τη δική μας την πλευρά. Ελπίζουμε να σταθούμε στο ύψος των προσδοκιών σας. Τώρα ο κύριο Ντερόι, ο οποίος είναι ε, νομικό, σύμβουλος επικρατεία για το Βέλγιο και επιστημονικός ε, συνεργάτης στο Πανεπιστήμιο τη Λουβέν. Έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ο χρόνος είναι περιορισμένος. Γι' αυτό και στην παρουσίασή μου θέλω να επικεντρωθώ στο άρθρο 44 της πρότασης οδηγίας εδώ κάποιες παρατηρήσεις από ε, μία εντάχει ανάγνωση της διάταξης δεν μπορεί παρά να είναι σημαντικές. Το άρθρο αυτό έχει τίτλο ε, «Δημόσιος έλεγχος». Σκοπό έχει να θεσπίσει έναν εξάρτητο, ενιαίο όργανο σε κάθε κράτος μέλος που να αναλαμβάνει τον έλεγχο και τον συντονισμό των δραστηριοτήτων ε, της υλοποίησης. Εν είδη εισαγωγής θα ξεκινήσουμε από την εξή ε, υπόθεση ότι ο έλεγχος υλοποίησης των οδηγιών για την ε, ανάθεση και την εκτέλεση των δημοσίων διαγωνισμών πραγματικά ευνοούν το συμβασμό των κανόνων αυτών. Πρώτα απ' όλα για δύο λόγους. Ο φόβος των ε, κυρώσεων που μπορεί να επιβάλλουν οι αρχές ή οι οποιασδήποτε παραβιάσεις. Φόβος που θα επηρεάσει τους συμμετέχοντες στην σχολαστική εφαρμογή των κανόνων. Δεύτερον, η σημασία της παρουσίας του ελέγχου αυτού είναι ότι η διαφήμιση, η διάδοση των αποτελεσμάτων του ελέγχου επιτρέπει ακριβώς να προσελκυστεί η προσοχή ε, στις διευθυντικές ε, δυσκολίες, στις συστημικές ε, ε, δυσκολίες που μπορεί να προκύπτουν λόγω της εφαρμογής των κανόνων. Έτσι μπορεί να γίνει μια, ε, επιτρέπουν να γίνεται μια νόμ, μόνιμη νομική παρακολούθηση των νομικών διατάξεων. Η σημασία λοιπόν του οργάνου αυτού θα πρέπει να οδηγεί σε αποτελεσματικούς έλεγχους, όπως αυτοί που προτείνονται από το άρθρο 44. Τουλάχιστον αυτό φαίνεται πρώτη όψεω να είναι ο στόχο. Ο μοναδικό χαρακτήρα του ενίου αυτού οργάνου που προτείνει η πρόταση οδηγία θα προσφέρει εγγύησει ε, για να αντιμετωπιστούν οι βασικέ δυσκολίε προσαρμογή. Σε καμία περίπτωση όμω δεν πρέπει να ξεχνούμε δύο σημαντικά στοιχεία, στα οποία θέλω να σταθώ. Πρώτον, υπάρχουν ήδη στο επίπεδο των διαφόρων κρατών μελών της Ένωσης συγκεκριμένοι μηχανισμοί ελέγχου που λειτουργούν και έχουν ανατεθεί σε αρμόδιες αρχές από καιρό μάλιστα. Δεύτερον, πρέπει να διερωτηθούμε για την διάρθρωση του ρόλου και του τρόπου που λειτουργούν τα διάφορα όργανα, το ενιαίο όργανο ελέγχου όπως προτείνεται και οι υπόλοιποι φορείς που ενδεχομένως ήδη να υπάρχουν. Δεύτερο σημείο, στο οποίο θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, είναι να δούμε κατά πόσον ο έλεγχος που διοργανώνεται βάσει των ε, μέτρων που προτείνονται στο άρθρο 44 δεν προκαλέσει τελικά δυσανάλογες συνέπειες. Στο έγγραφο εργασίας που θα σας υποβληθεί προσεχώς, εφόσον ολοκληρωθεί, Αναφέρω ανακεφαλαιωτικά και ενίδη παραδείγματο κάποιε μορφέ ελέγχου όπω έχουν ε, προταθεί στο Βέλγιο. Διοικητικού ελέγχου, ελέγχου δικαιοδοσία και πολιτικού ελέγχου. Ε, η σημασία τη σύνοψη αυτή τώρα για τι μορφέ ελέγχου είναι η εξή. Θέλουμε να ε, παρατηρήσουμε ότι όσο και αν είναι ποικίλη η έλεγχη αυτή, τελικά είναι αρκετά διαδεδομένη παρόλα αυτά δεν καλύπτουν αναγκαστικά το σύνολο των πρακτικών σε σχέση με τους δημόσιους διαγωνισμούς. Ιδανικά ένα ενιαίο μοναδικό εργαλείο θα επιτρέπει να υπάρξει προστιθέμενη αξία ως προς τις ε, περιοχές όπου δραστηριοποιούνται οι δημόσιοι διαγωνισμοί και αυτή τη στιγμή δεν φωτίζονται από την, ε, το φως ακριβώς του ελέγχου. Θέλω να σταθώ επίσης σε άλλα δύο σημεία. Η διάρθρωση του ρόλου και του τρόπου δράσης των ε, ε, μοναδικών των ενιαίων εργαλείων ε, ελέγχου και των υπόλοιπων φορέων που είναι αποφορτισμένοι με τον έλεγχο των διαδικασιών δημοσίων διαγωνισμών. Ε, Σύντομε παρατηρήσει, γιατί σα παραπέμπω και στο έγγραφο το οποίο σα ε, ανέφερα προηγουμένω. Κάποιε παρατηρήσει που μου εμπνέει η ανάγνωση του άρθρου 84, σημείο 3 τη οδηγία. Το σημείο Α παρακολούθηση των κανόνων που έχουν να κάνουν με τις δημόσιες προμήθειες. Έλεγχο που έχει αναλάβει ακριβώς το ενίο εργαλείο ελέγχου. Η παρακολούθηση αυτή θα πρέπει να είναι συστηματική ή να διεξαγάγεται όταν υπάρχουν έκτακτες ε, περιστάσεις, λόγω χάρη προσφυγή. Η διάκριση μεταξύ της παρακολούθησης όπως αναφέρεται στο σημείο Α και της αρμοδιότητας ε, ε, εξέτασης προσφυγές προσφυγών, όπως αναφέρονται στο σημείο 3 ΣΥΓΜΑΤΑΦ, αυτή η διάκριση δεν είναι σαφή. Το άρθρο 84.3 Β αναφέρει ότι το όργανο αυτό είναι επιφορτισμένο με δικαστική αρμοδιότητα ε, ανάθεσης. Το πρώτο ερώτημα που έρχεται στο νου είναι πόσο το όργανο αυτό έχει αρμοδιότητες τέτοιες ελέγχου και ανάθεσης παράλληλες, ώστε να μην υπάρχει και ασύμβατο. Δηλαδή, ο έλεγχος ανατίθεται σε ένα όργανο το οποίο προχωράει σε διαβουλεύσεις ή μπορεί να γνωμοδοτεί. Στο σημείο 84.3 ε υπάρχει η αρμοδιότητα να επισημαίνεται στις εθνικές αρχές, ιδίω τις αρχές ε, ελέγχου, αν υπάρχουν παραβιάσεις συστηματικές ή συστημικές. Και πάλι προκαλείται σύγχυση από το κείμενο. Μεταξύ των δυνατοτήτων ε, προσφυγή σε δικαιοδοσία, των αρμοδιοτήτων ελέγχου και το τι ε, δρόμο θα πάρουν τελικά οι προσφυγές βάσει τις οδηγίες όπως προτείνεται. Το σημείο 84 84-3 σιγματάφ επιφορτίζει το εθνικό αυτό όργανο ελέγχου με την εξέταση των προσφυγών πολιτών και επιχειρήσεων σε ό,τι αφορά την υλοποίηση των κανόνων σε σχέση με του δημόσιου διαγωνισμού. Εδώ το πρόβλημα είναι ότι δεν αντιλαμβάνεται κανεί ε, με μια πρώτη ανάγνωση κειμένου και πρώτη όψεω πώ διαρθρώνονται αυτή η εξέταση των προσφυγών από τη μια και οι προσφυγές ε, σε δικαιοδοσίε από τις επιχειρήσεις κατά τα άλλα. Η αρμοδιότητα αυτή μας θυμίζει και την πιθανότητα ασυμβάτου μεταξύ της αρμοδιότητας παρακολούθησης και ελέγχου. Τώρα στο σημείο 84 3 εδώ αναφέρεται η αρμοδιότητα του οργάνου να εξετάζει και προδικαστικά κάποιες υποθέσεις ή εφόσον αποφανθεί το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο. Τι εννοούμε τελικά με τον έλεγχο, ότι θα εξασφαλίζεται η συμβατότητα των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, γιατί σε αυτή την περίπτωση δεν ξέρουμε αν χρειάζεται πραγματική ανάθεση ευθύνη ή θα εξασφαλίσετε συνέχιση των αποφάσεων που θα λαμβάνουν οι εθνικέ δικαιοδοσίε, τα εθνικά δικαστήρια. σω ένα τέτοιο σύστημα προκαλεί και άλλε πιθανότητε ασυμβάτου. Ε, ουσιαστικά προκαλώντας σύγχυση στις αρμοδιότητες δικαιοδοσίες ε, των εθνικών οργάνων, των εθνικών φορέων. Πώς μπορεί μια διοικητική αρχή να ελέγχει τις αποφάσεις ε, των εθνικών δικαιοδοσιών. Τώρα, για το 84-4 αναφέρονται κάποιες υποχρεώσεις που μπορεί να επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο όργανο ελέγχου. Εδώ πρέπει κανείς να διασφαλίζει ότι η υποχρεώσει αυτέ εκπληρώνονται με τρόπο συμβατό με αυτόν που πρέπει να λειτουργούν και οι εθνικές αρχές. Τώρα, ένα δεύτερο σημείο το οποίο θέλω να θίξω σύντομα, γιατί και αυτό τράβηξε την προσοχή μου κατά την ανάγνωση του άρθρου 84, είναι ο αναλογικός χαρακτήρας των ελέγχων και τη αποστολή που έχει αναλάβει αυτό το εθνικό όργανο. Σε γενικέ γραμμέ, μπορεί να αναρωτηθεί κανεί, εάν η διοργάνωση αποστολών ελέγχου εφόσον μάλιστα ο έλεγχος εγγράφεται στη διαδικασία ανάθεσης. Μπορεί κανείς να ρωτηθεί εάν τέτοιοι έλεγχοι δεν επιβαρύνουν δυσανάλογα τελικά την διεξαγωγή της διαδικασίας ανάθεσης συμβάσεων. Μπορεί επίσης κανείς να διερωτηθεί κατά πόσον η διοργάνωση των ελέγχων αυτών δεν περιπλέκει έτσι περαιτέρω το σύστημα. Και θα συμφωνήσω εδώ με τη συνάδελφο, την κυρία ε, Μέγκελε, που εξέφρασε παρόμοιε ανησυχίε. Και εδώ το συμπεράσμά μου, καθότι ο χρόνο που μου έχει διατεθεί θα λήξει. Σε γενικέ γραμμέ, ο αποτελεσματικό έλεγχο θεωρείται ένα στόχο προφανώ επενεταίο και θεμητός αλλά από τις διατάξεις του άρθρου 84 της οδηγίας προκαλούνται ανησυχίες, προκαλούνται φόβοι ότι ο θεσμός ενός τέτοιου οργάνου δεν συνδυάζεται αρμονικά με τους προϋπάρχοντες μηχανισμούς στα διάφορα κατημέλη. Μπορεί λοιπόν κανείς να αναρωτηθεί για την ε, σχέση κόστους-οφελίας, πρόβλεψης ενός τέτοιου συστήματος ελέγχου, εφόσον ε, Μιλάμε για διαδικασίε που μπορεί να βρισκόνται και σε εξέλιξη. Δεν θα πρέπει οι υπέρμετροι έλεγχοι να βλάπτουν τον ίδιο τον έλεγχο. Σα ευχαριστώ. Well, thank you very... Και εμεί σα ευχαριστούμε. Κοίταζα το 84 όσο μιλούσατε και συμμερίζομαι τις ανησυχίες σας. Ίσως ο εισηγητής μας επανέλθει σε αυτό αργότερα. Τώρα για κάτι πιο θετικό. Οι πιο καινοτόμες προμήθειες ενδιέφεραν και τον εισηγητή μας για το θέμα του 6, του 2006. Ο επόμενος εμπειρογνώμων, Κριστόφ Βέης, είναι ακριβώς ειδικό για το θέμα προμήθειες και καινοτομία. Με μεγάλη χαρά του δίνω το λόγο για 10 ολόκληρα λεπτά για να αξιολογήσει τις προτάσεις της Κομισιόν στο θέμα της καινοτομία. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, καταρχήν ευχαριστώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την πρόσκλησή του για να δώσουμε την άποψή μας για την καινοτομία στη νέα πρόταση. Είμαι από την υπηρεσία καινοτομία της φλαμανδικής κυβέρνησης που δημιουργήθηκε το 9 μετά από απόφαση της φλαμανδικής κυβέρνησης mm. και το πρώτο μας θέμα ήταν η δημιουργία ενός κέντρου γνώσης για τις προμήθειες και μετά προσπαθήσαμε να δούμε ποια μεθοδολογία είναι η καλύτερη για το PPI και το PCP. Μέχρι τώρα εξετάσαμε πολλά πιλωτικά προγράμματα και η φλαμανδική κυβέρνηση ενέκρινε 10 εκατομμύρια για τα πιλωτικά αυτά προγράμματα. Στη διαφάνεια αυτή βλέπετε τι ισχύει στην Ευρώπη Μόνο τρεις χώρες εφαρμόζουν όσα έχουμε συζητήσει. Δηλαδή όλες οι άλλες χώρες αρχίζουν μόλις να ταυτίζουν πιθανά πιλωτικά προγράμματα για τη βελτίωση των προμηθειών. Το θέμα μπορεί να τεθεί λοιπόν το ερώτημα είναι πολύπλοκες οι οδηγίες και πρέπει να απλοποιηθούν. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο διστάζουν οι χώρες μέλη να εφαρμόσουν τα συμπεφωνημένα δηλαδή να εφαρμόσουν πιλωτικά πειραματικά προγράμματα. Κάτι εμάς θα έπρεπε να καλύψουμε δύο κατηγορίες. Πρώτον, που μάλιστα ξεχνιέται συνήθως, είναι η προμήθεια καινοτόμων λύσεων αγαθών και υπηρεσιών Μπορεί να είναι νέες καινούριε για το ένα συμβαλόμενο μέρος, αλλά υπάρχουν ήδη στην αγορά. Και η άλλη κατηγορία είναι η αγορά καινοτόμων προϊόντων, υπηρεσιών ή διαδικασιών που δεν υπάρχουν ακόμη στο, στην αγορά με στόχο να λύσουν κοινωνικο-οικονομικά προβλήματα και να βελτιώσουν τη λειτουργικότητα των δημοσίων υπηρεσιών. Σήμερα η καινοτομία στον τομέα των δημοσίων προμηθειών θεωρείται κάτι πολύ εύκολο. Εκτός από την ε, προσαρμογή της νομοθεσίας απαιτείται και μία αλλαγή νοοτηροπίας και δεν νοείται παρά μόνο αν όσοι λαμβάνουν τις αποφάσεις είναι διατεθειμένοι να δουν τα πράγματα όπως είναι. Η δημόσια προμήθεια καινοτομίας απαιτεί καταρχήν πολλούς εμπειρογνώμονες Δεν μπορούν μόνες τους οι αρχές να τα λύσουν όλα. Γι' αυτό χρειάζονται εμπειρογνώμονες, ειδικοί στις προμήθειες, στην καινοτομία, που γνωρίζουν δηλαδή τεχνικά τα πράγματα για να κάνουν την απαραίτητη αξιολόγηση των καινοτομιών. Επίσης χρειάζονται πολλές φάσεις και αυτό λείπει στην τωρινή πρόταση. Με βάση την εμπειρία μας Νομίζουμε ότι για να μιλήσουμε για καινοτομία χρειάζονται τρεις φάσεις. Πρώτον, ομαδοποίηση των, της ζήτησης. Για να μπορέσουμε να κάνουμε αξιολόγηση της κατάστασης και να δούμε πώς να προωθήσουμε την καινοτομία. Δεύτερη φάση, προεμπορική προμήθεια. δηλαδή δημιουργία πρωτοτύπων για να επιτρέψει αυτό στις αρχές να εξετάσουν κατά πόσον αυτά που θέλουν να αγοράσουν ή να προμηθευτούν είναι χρήσιμα σύμφωνα με το πρωτότυπο. Και η τρίτη φάση βέβαια είναι η κανονική, ο κανονικός διαγωνισμός. Τώρα, για την προτινόμενη οδηγία. Άκουσα πολλούς να μιλάνε για καταστροφή. Εγώ εμείς νομίζουμε ότι η απλοποίηση είναι κάτι που πρέπει να προβλεφθεί. Είπατε κύριε Χάρμπορ ότι η πρόταση τονίζει τη σημασία των δημοσίων προμηθειών για την καινοτομία και ότι πρέπει να παίξει σημαντικό ρόλο και σημαντικότερο ακόμη στο μέλλον. Η έρευνα και η καινοτομία είναι η κύρια ορμή για την επίτευξη των στόχων του 2020. Παρ' όλα αυτά, με την προτινόμενη οδηγία υπάρχουν και ορισμένες, η προτινόμενη οδηγία δημιουργεί και ορισμένες ανησυχίες. Για να ενθαρρύνουμε τους προμηθευτές και προμηθεύτριες να χρησιμοποιήσουν αυτό το εργαλείο όπως πρέπει. υπάρχει ένα σαφές πρόβλημα, ένας διαχωρισμός που πρέπει να γίνει μεταξύ των διαφόρων δυνατοτήτων που δίνει η πρόταση. Πρώτον, ο αποκλεισμός του άρθρου 13 για τις υπηρεσίες στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης και έπειτα χωριστά οι καθεαυτού διαδικασίες προμηθειών. Αν πράγματι υπάρχει θέληση να προμηθευτούν οι αρχές καινοτόμες υπηρεσίες και αγαθά, πρέπει να γνωρίζουν ποια διαδικασία πρέπει να ακολουθήσουν. Η σαφήνεια λοιπόν είναι κάτι τελείως απαραίτητο. Οι προμηθευτές και προμηθεύτριες δεν είναι ειδικοί στον τομέα της καινοτομίας. Άλλο πρόβλημα είναι ότι η έννοια της έρευνας και ανάπτυξης R&D δεν είναι σαφής. Για την άμυνα ας πούμε είναι σαφές το γιατί δεν υπάρχει ο ίδιος ορισμός Uh, Όπως και για το GPA. Uh, Ένα άλλο πρόγραμμα που θέλω να αναφέρω βρίσκεται στο προήμιο στην εισαγωγή της πρότασης όπου γίνεται παραπομπή σε καινοτόμες εταιρικέ σχέσεις και τίποτε άλλο. Ούτε το PCP ούτε το R&D. Επομένως, κανείς δεν είναι διατεθειμένος να εγκρίνει νέες διαδικασίες αν δεν υπάρχει σαφής αναφορά στο νομικό υπόβαθρο που ισχύει παράδειγμα ως μία από τις πρώτες χώρες στην Ευρώπη που άρχισαν το πρώτο πρόγραμμα PCP οι αρχές δεν βρήκαν σαφή νομική βάση ή υπόβαθρο στην ισχύουσα νομοθεσία για την εφαρμογή του PCP. Παρόλα αυτά, τώρα ζητήσαμε από την Κομισιό να αποσαφηνίσει τους κανόνες για να μπορούν τα κράτη-μέλη που θέλουν να ακολουθήσουν τέτοια διαδικασία να την ακολουθήσουν. Άλλο πρόβλημα που υπάρχει στην πρόταση αφορά το IPR που αναφέρεται μεν ρητά αλλά χωρίς καμία κατευθυντήρια γραμμή για το πώς θα εφαρμόζεται. Πρέπει να αποσαφινιστούν όλα αυτά λοιπόν και για τα πνευματικά δικαιώματα. Επίσης για τις κοινέ διαμεθοριακές προμήθειες προβλέπετε κάτι αλλά το οποίο αντιφάσκει με την ιδέα, με την ιδέα του μοιράσματο των συμβολέων που προτείνεται. Αν συνδυάσουμε τη ζήτηση που αυξάνεται με την πρόταση θα καταλάβουμε γιατί οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν είναι πρόθυμες να την εφαρμόσουν. Η αποσαφήνιση λοιπόν της χρήσης της διαδικασίας αυτής χωρίς δημοσίευση για τις προμήθειες καινοτόμων προϊόντων είναι κάτι που λείπει. Για τις καινοτόμες εταιρικέ σχέσεις, για τις εταιρικέ σχέσεις καινοτομίας. Είναι κάτι που μοιάζει με το forward commitment procurement προφανώς. Πώς μπορεί να εφαρμοστεί μια τέτοια διαδικασία και να καταλήξει στην προμήθεια. Το πρόβλημα είναι ότι όταν υπάρχει ένα συμβόλαιο με κάποιον προμηθευτή, μακροχρόνιο μάλιστα, τελικά προωθούνται οι μεγάλες επιχειρήσεις αντί των μικρομεσαίων. Υπάρχει και ένα πρόβλημα διπλής χρηματοδότησης. Θέλουμε οι προμηθευτές να έχουν τα πνευματικά δικαιώματα που δικαιούνται, αλλά δεν είμαστε βέβαιοι ότι θα δεχτούν τις νέες αυτές διαδικασίες, γιατί δεν είναι φανερό σε κατά τι διαφέρουν με τη γνωστή συνήθη διαδικασία του PCP. Παραμένουν αυτά τα προβλήματα. Τώρα θα ήθελα για να τελειώσω. Υπάρχει η δυνατότητα στα πλαίσια του προγράμματος 2020 να τονίσουμε έναν προϋπολογισμό που να προωθεί τις βέλτιστες πρακτικές και την καινοτομία στην Ένωση. Οι προμηθευτές και προμηθεύτριες σήμερα αναγκάζονται να προμηθεύουν με πρασινότερο λέει τρόπο και πιο καινοτόμο. Αλλά πώς να μην συγχέσουν όλα αυτά τα πράγματα στο μυαλό τους. Πολύ δύσκολο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας έδωσα λίγο περισσότερο χρόνο γιατί με ενδιαφέρουν ιδιαίτερα τα θέματα αυτά. Αυτό που μας λέτε όμως είναι ότι η Κομισιόν πρέπει να λειτουργήσει καλύτερα, να προσπαθήσει περισσότερα, συμμεριζόμαστε το στόχο, αλλά πρέπει να εργαστεί περισσότερο. Και ο τελευταίος μας εμπειρογνώμων μιλάει για νέες τάσεις και νέα εργαλεία. Ο Πάολο Μαζίνια, ο οποίος είναι ο πρόεδρος της Εθνικής Υπηρεσίας Προμηθειών στην Πορτογαλία και η Πορτογαλία ήταν ένας από τις ηγέτες της Ευρώπης σε ηλεκτρονικές προμήθειες. Χαίρομαστε ιδιαίτερα που θα σας δώσουμε το λόγο για 10 όμως λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, κύριε Συγητή, μέλη της Επιτροπής. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είναι τιμή μου και μεγάλη χαρά να βρίσκομαι εδώ σήμερα. Σε αυτή την ακρόαση. Πιστεύω ότι καλύτερα από τα λόγια ή είχε και εικόνες είναι πιο αποτελεσματική. Γι' αυτό θα σας προσκαλέσω να δείτε το βίντεο.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 The challenge is to promote interoperability, e-signatures, e-authentication and e-identification mechanisms, which can only be achieved through collaboration between all member states. Portugal is ready for that challenge. Well, thank you. Well, thank Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε που κάπως κάνατε πιο χαρούμενο το απόγευμά μας. Θα ήθελα βέβαια κάποια πράγματα να τα εξηγήσω, αν μου επιτρέπετε. Ελπίζω να το στείλατε αυτό και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην αρχή της μελέτης τους, έτσι. Ναι. Αυτή ήταν η ιδέα του τμήματος ε, των δημιουργών. Δεν φταίω εγώ γι' αυτό. Ούτε για το πράσινο. Τέλος πάντων, οι ηλεκτρονικές ε, προμήθειες είναι στα πλαίσια της ε, ατζέντα της Ευρώπης για το 2020 για να έχουμε μεγαλύτερη ανάπτυξη και απασχόληση μεταξύ άλλων. Νομίζω θα μπορούσαμε να υποφεληθούμε από το παράδειγμα της Πορτογαλίας, τις ηλεκτρονικές δημόσιες προμήθειες. Εμείς τα καταφέραμε και νομίζω ότι μπορούμε να βελτιώσουμε τη διαδικασία δημοσίων διαγωνισμών εποφελούμενοι και από τις ε, διαφορετικές τάσεις. Νομίζω, νομίζω ότι οι τάσεις λοιπόν στον τομέα IT θα μπορούσαν να επιτρέψουν τον εξορθολογισμό πόρων στις δημόσιες αρχές με τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες, την ανταγωνιστικότητα και την προσφορά περισσότερων λύσεων. Η ε, ηλεκτρονική διαδικασία ήταν φυσική επιλογή στα πλαίσια ευρύτερης μεταρρύθμισης που ξεκίνησε το 2007 στη χώρα μας. Στόχος ήταν να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα των δημοσίων αρχών και υπηρεσιών. Βεβαίως, η δημιουργία της υπηρεσίας, ο κεντρικός χαρακτήρας των αγορών και η δημιουργία ενός ενιαίου μοντέλου ήταν ε, αποφασιστικά εργαλεία για να δημιουργήσουμε ένα σύστημα βιώσιμο. Ε, καταφέραμε να συγκεντρώσουμε όλους τους ε, βασικούς ενδιαφερομένους στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και έτσι επιφέραμε τις αλλαγές που απαιτούνταν ώστε να υπάρξει και απαραίτητη πολιτική εφαρμογή. Σε αυτό το πλαίσιο, ε, οι ηλεκτρονικές δημόσιες προμήθειες επέτρεψαν να μετατοπιστούμε από το παραδοσιακό μοντέλο σε ένα στρατηγικό εργαλείο, ώστε να έχουμε περισσότερα και καλύτερα αποτελέσματα. Η χρήση της ηλεκτρονικής οδού από, τον, ε, από το 2009 είναι υποχρεωτική στην Πορτογαλία. Νομίζω κανένα δημοσιοέργο δεν ανεστάλλει, δεν διακόπει για το λόγο αυτό καμία παράδοση αγαθού ή εμπορεύματο ε, ή υπηρεσία δεν ε, ανεβλήθη λόγω αυτής της διαδικασία. Απλώ προσαρμόσαμε το νομικό μας πλαίσιο. Κάτι που μας επέτρεψε το, το κατά πρώτη όψη εκρηκτικό μείγμα των πολιτικών ηθινόντων, των ε, μάνατζερ, των δημιουργικών υπηρεσιών και αν δεν το πιστεύετε και των δικηγόρων. Έτσι, συνδυάσαμε τη ζήτηση με την αποκέντρωση. Ήταν σαφής η δέσμευση όλων των συμμετεχόντων, ιδιωτών και δημοσίων. Οι πλατφόρμες ε, των ηλεκτρονικών διαγωνισμών μάλιστα αυτή τη στιγμή είναι στα χέρια ιδιωτών ήδη. Μιλάμε για μια κατάσταση που αποφέρει κέρδη σε όλους, και την κυβέρνηση και τις ε, επιχειρήσεις και τις συμβάλλουσες αρχές και τις φορές τοπικής αυτοδιοίκησης. Αγορές ανοίγουν σε νέους οικονομικούς φορείς, και εμπορευμένου, ιδίω στι μικρομεσαίε επιχειρήσει. Ο ανταγωνισμό και η ανταγωνιστικότητα τονώθηκαν. Πετύχαμε μεγάλε εξοικονομήσει. Η διαφάνεια και η ευκολότερη πρόσβαση πραγματικά είναι, προόδευσαν. Όμω, ω τώρα επικεντρωθήκαμε στου ηλεκτρονικού διαγωνισμούς καταλάβαμε ότι μόνο εάν η ηλεκτρονική εδώ καλύπτει όλη την αλυσίδα του διαγωνισμού μπορούμε να παρακολουθήσουμε σε μεγαλύτερη κλίμακα από άποψης άποψη το τι μπορούμε να πετύχουμε με τους δημόσιους διαγωνισμούς. Με το ηλεκτρονικό μας μοντέλο θα πετύχουμε, πιστεύουμε, τρεις ε, βασικούς στόχους. Οικονομικούς, κοινωνικούς και πολιτικούς. Από οικονομικής άποψης θα έχουμε μεγαλύτερη εξοικονόμηση κονδυλίων και θα μειώσουμε τις δημόσιες δαπάνες κοινωνικός, επειδή θα παρέχουμε καλύτερε υπηρεσίε προ του ενδιαφερομένους και θα βελτιωθεί η λειτουργία των δημοσίων αρχών. Λαμβάνοντα υπόψη και τα σχόλια των προηγούμενων εμπειρογνωμόνων. Και από πολιτική άποψη, με διαφανή, αυστηρό και αποτελεσματικό τρόπο διεξαγωγή των διαγωνισμών. Θα υπάρχει περισσότερη λογοδοσία και μεγαλύτερη απόδοση πτυνών. Άρα, Προσωπικώ πιστεύω ότι η ηλεκτρονική οδό για του δημόσιου διαγωνισμού θα μα επιτρέψει να δημιουργήσουμε ένα νέο μοντέλο στην ε, δημόσια διοίκηση. Περνώντα από τα απλά εργαλεία IT σε μια πραγματικά ηλεκτρονική στρατηγική δημοσίων συμβάσεων. Και θα δημιουργηθεί ένα ε, κοινό ε, επίση ίσης και βιώσιμο εργαλείο, ώστε να κινηθούμε αποτελεσματικά στον χώρο των δημοσίων πολιτικών, ιδίω προ του δημόσιου διαγωνισμού. Αγαπητέ Πρόεδρε, μέλη της Επιτροπής, θα ήθελα να ολοκληρώσω παρουσιάζοντας κάποιες από τις απόψεις μας σε σχέση με την ηλεκτρονική διεξαγωγή ε, δημοσίων διαγωνισμών. Η χρήση των νέων, καινοτόμων και ισχυρών εργαλείων θα πρέπει να επιτρέπει και αλλαγές στην όλη αλυσίδα. Θα πρέπει να αφιερώσουμε χρόνο και προσπάθειες σε ένα σφαιρικό μοντέλο ηλεκτρονικών διαγωνισμών, ώστε να υπάρχει αξιοπιστία, εμπιστοσύνη, υψηλές δεξιότητες, και διαφάνεια. Θα πρέπει με γνώσεις και δεξιότητα να διασφαλίσουμε αυτά που θέλουν οι ενδιαφερόμενοι και οι φορολογούμενοι. Τα κράτη-μέλη μπορούν να χρησιμοποιήσουν τους ηλεκτρονικούς διαγωνισμού, αλλά δεν πρέπει να παραμείνουμε σε αυτή τη δήλωση. Θα, ε, θα μπορούσαν να χρησιμοποιούν την ηλεκτρονική οδό τα κράτη-μέλη. Αυτό ελπίζουμε το λάβει υπόψη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την ευκαιρία της αναθεώρησης ε, των οδηγιών. Ε, νομίζω ότι έλειξε ο χρόνος. Με ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος, για την υποστήριξη όλης αυτής της διαδικασίας. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η σειρά των παρουσιάσεων των εμπειρογνωμόνων. <clears throat> Τώρα κάπως ξεπερνάμε το χρόνο μας, αλλά ήθελα να δώσω στα μέλη της Επιτροπής μας να κάνουν κάποια σύντομα σχόλια αν θέλουν. Κυρία Βάιλερ, κυρία Ρούλε, ποιος άλλος θα ήθελε να θέσει ερωτήματα για το δεύτερο γύρο. Βάιλερ, Ρίλε, όποιος άλλος θέλει να λάβει το λόγο, ευχαριστώ. Κύριε Βάιλερ πρώτα, για ένα λεπτό, <coughs> αν δεν σας πειράζει. Κύριε Πρόεδρε, ήταν ενδιαφέρουσα και εντυπωσιακή η η τελευταία παρουσίαση μετά τις πολλές επικρίσεις που είχαμε ακούσει. Ίσως ε, ήταν πάρα πολλοί οι νομομαθείς από τη Γαλλία και τη Γερμανία που επεξεργάστηκαν την πρόταση της Κομισιόν και πολύ λίγοι από την Πορτογαλία που θα την κάναν πολύ πιο ελαφρότερη την πρόταση. Εγώ και από τη δική μου πολιτική ομάδα συμμερίζομαι την άποψη ότι έχουμε ζητήσει ίσως πάρα πολλά από την νομοθεσία, αλλά όλα αυτά μπορούν να τροποποιηθούν. Έχω ένα ερώτημα τώρα. Στον προηγούμενο ομιλητή, τον κύριο Κρίστοφ Βάις, είπατε κι εσείς κάτι το οποίο το βρήκα πολύ σημαντικό, πέρα από τα κοινωνικά κριτήρια, αναφερθήκατε στο θέμα της έρευνας και της ανάπτυξης. Ε, από ό,τι βλέπω εδώ πέρα στις διαφάνειές σας, αναφερθήκατε ότι δεν μπορεί να υπάρξει το λεγόμενο double founding για τα συστήματα πληροφορικής βάσει των τωρινών κανόνων. Ε, συμπεραίνω σωστά ότι δεν μπορεί κανείς να ε, αλλάξει αυτό το πράγμα. Τι ακριβώς εννοείται τώρα στο double founding, θα ήθελα να ξέρω. Είναι ίσως μια πρόσθετη επιλογή, αλλά χωρίς να δίνονται προνόμια σε κάποιους. Θα ήθελα να μου εξηγήσετε τι ακριβώς εννοείται με το double founding. Ευχαριστώ κύριε Αριούλη, ευχαριστώ πολύ. Και εγώ θέλω να ευχαριστήσω τους ομιλητές και για τον κύριο Βάις θα ήθελα να θέσω ορισμένα λεπτομεριακά ερωτήματα. Δεν θέλω όμως τώρα αυτό να το συζητήσω, να μου απαντήσει. Περισσότερο με την κυρία Μάισνερ θέλω να στραφώ. Το άρθρο 11 για, το, για τη συνεργασία μεταξύ δημόσιων τομέων. Και τώρα έρχομαι στο θέμα του ανταγωνισμού. Στη Γερμανία υπάρχει μια κάτι το οποίο είναι δύσκολο να μεταφράσει κανείς. Προσπαθούμε με ένα φορέα μονάχα να έχουμε οικονομικό, τεχνικό και ε, νομικό έλεγχο. Εμείς, εγώ θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει διαφορετική εποπτεία οι πολιτικές αρχές, τον πολιτικό έλεγχο, τον νομικό έλεγχο, οι δικαστικές αρχές και τον οικονομικό, το ελεκτικό συνέδριο. Είναι πολύ δύσκολο λοιπόν να φέρει κανείς αυτά τα θέματα από κοινού και γι' αυτό ήθελα να θα σας θέσω αυτό το ερώτημα. Μετά το άρθρο 11 για τις συνεργασίες δημόσιου τομέα με δημόσιο τομέα. Θέλετε ότι αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη στην οδηγία το ή όχι. Εγώ το πρόβλημα είναι να μην αποκλειστεί επειδή δεν αναφέρεται κάτι τέτοιο. Νομίζω ότι η συνεργασία σε οριζόντιο και νότιο <coughs> και κάθε το επίπεδο μεταξύ δημοσίων φορέων θα πρέπει να επιτρέπονται μέσα στα πλαίσια της ε, αυτοδιοίκησης των τοπικών και περιφερειακών τομέων και εδώ δεν βλέπω να αναφέρονται στην οδηγία της Κομισιόν. Εγώ νομίζω ότι αυτό είναι απαραίτητο να αντιμετωπιστεί από αυτήν την οδηγία γιατί είχαμε πολλές νομικές διαμάχες στο παρελθόν και θα πρέπει εδώ να υπάρξει και κάποια διευκρίνηση. Ευχαριστώ. Δίνω το δύο λεπτά στο κάθε από τους εμπειρογνώμονες. Δεν ξέρω κάποιο άλλο μέλος αν θέλει να θέσει ένα ερώτημα. Εντάξει. Ας ξεκινήσουμε και πάλι ανάστροφα. Ο κύριος Μεζίνα πρώτος ε, θα απαντήσει ή μπορεί να μας δώσει κάποιο μήνυμα αν θέλει πέραν του, της υποστήριξης του, της των ηλεκτρονικών προμηθειών που παρουσίασε προηγουμένω. Και μετά γυρίζουμε με αναστροφή σειρά στου άλλου ομιλητέ. Κύριε Μαζίνα. Το μήνυμά μου είναι πολύ σαφέ. Έχουμε αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο ακούμε μουσική, έχουμε αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο διαβάζουμε. Γιατί να μην αλλάξουμε και τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε τι δημόσιε προμήθειε. Η ιδέα μα είναι να θέσουμε σαν πρότυπο το e-procurement, τι ηλεκτρονικέ προμήθειε και μετά να εφαρμόσουμε τις αρχές της συνθήκης. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλος τρόπος να το πετύχουμε αυτό για να δώσουμε καλύτερη χρήση στις δημόσιες, ε, να είναι πιο χρήσιμες οι δημόσιες προμήθειες. Κύριε Βέης, εσείς νομίζω ήσασταν το αντικείμενο των περισσότερων ερωτήσεων για το λεγόμενο double funding. Για το double funding που είναι διπλή χρηματοδότηση τελικά, όχι διπλή ίδρυση. Αν μια εταιρεία συμμετέχει σε μια καινοτόμα διαδικασία σε μια χώρα για ένα συγκεκριμένο θέμα και παίρνει χρηματοδότηση, αν θέλετε να το πείτε αυτό, τότε δεν μπορεί να συμμετάσχει σε ένα άλλο κράτος μέλος σε αντίστοιχη χρηματοδότηση για καινοτόμες διαδικασίες για το ίδιο θέμα. Επειδή θεωρείται ότι έχει ήδη πάρει χρηματοδότηση με την πρώτη διαδικασία σε ένα άλλο κράτος μέλος. Αυτό είναι το double funding, όχι founding, για την διπλή χρηματοδότηση κατά κάποιο τρόπο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ντερόι. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να απαντήσω στο ερώτημα το οποίο έθεσε η κυρία Ρίλε. Πράγματι, το να δοθούν όλες οι μορφές ελέγχου, είτε είναι πολιτικός, είτε είναι νομικός, είτε είναι οικονομικός, σε ένα φορέα μονάχα, Επομένως, το να θέσουμε σε ένα μονάχα φορέα όλα αυτά τα, όλες αυτές τις μορφές ελέγχου, ετέθη το ερώτημα αν δημιουργεί προβλήματα. Δεν είναι πρόβλημα αν αυτό ήταν ο στόχος των συντακτών αυτής της ε, οδηγίας, γιατί κανονικά οι έλεγχοι έχουν διαφορετικό στόχο. Ο οικονομικός έλεγχος αφορά την χρήση των ε, δημοσίων κονδυλίων ένας νομικός έλεγχος έχει σαν στόχο να εξασφαλίσει την προστασία των επιχειρήσεων που θεωρούν ότι έχουν φύγει σε μια διαδικασία ή ακόμα και για να κολλάσει ποινικά ορισμένε συμπεριφορέ, οι οποίε επισύρουν μια δίωξη αν υπάρξει απάτη κτλ. Επομένω, το να δώσουμε όλε αυτέ τι ε, αρμοδιότητε σε ένα μονάχα φορέ, αυτό μπορεί να οδηγήσει πρόβλημα. Μα είναι αυτό η πρόθεση των συντακτών τη πρόταση αυτή, Εγώ, διαβάζοντα το άρθρο 84 δεν βλέπω να είναι σαφή τα πράγματα. Θα πρέπει να θεωρήσουμε ότι αυτό το ελεκτικό όργανο θα έχει μία υπολοιπόμενη αρμοδιότητα για να καλύψει τις, ε, τους ελέγχους που δεν κάνουν άλλοι φορείς και αυτό είναι μία <clears throat> δυνητική ερμηνεία. Θα μπορούσε κανείς να θεωρήσει ότι αυτό το εργαλείο έχει ένα ρόλο συμπληρωματικό και εξασφαλίζει τουλάχιστον την πλήρη κυκλοφορία των πληροφοριών μεταξύ όλων των παρεμβενόντων και τότε ο ρόλος του θα έδινε πραγματικά μια προσθέμενη αξία. Αλλά το να δώσουμε την εντύπωση ότι συγκεντρώνονται όλοι οι έλεγχοι σε ένα μονάχα όργανο, αν είναι ρεαλιστικό αυτό ή όχι, νομίζω ότι αυτό θα δημιουργήσει αρνητικές ε, αντιμετωπίσεις και θα θίξει το ρεαλισμό αυτής της πρότασης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Τέλος η κυρία Ποθ Μέγκελε, σας ευχαριστώ και εγώ για το θέμα του άρθρου που έχει να κάνει με τη διακυβέρνηση και το νέο θεσμό. Συμφωνώ σε αυτό που είπε η κυρία Ρούλε. Είναι όπως και η Βουλή της των Κοινοτήτων στο Ηνωμένο Βασίλειο που τόνισε ότι υπάρχουν ορισμένα θέματα τα οποία υπόκεινται στην ε, επικουρικότητα και πρέπει να γίνονται σε επίπεδο κρατών μελών. Σε ό,τι αφορά τη συνεργασία μεταξύ δημοσίων υπηρεσιών, εγώ είχα <clears throat> να διατυπώσω την πρόταση να υπάρξει μια προστίκη για το άρθρο 1 σε σχέση με το αντικείμενο που να συμπεριλάβει και αυτά τα στοιχεία τα οποία τα τόνισε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο ψηφισμά του αυτά μάλλον που απαρίθμησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως κριτήρια για να μπορέσει να υπάρξει συνεργασία μεταξύ δημοσίων αρχών. Να εξαιρεθεί λοιπόν σε αυτές τις περιπτώσεις η συνεργασία αυτή. Ευχαριστώ. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους πάρα πολύ και τους οκτώ τους εμπειρογνώμονές μας για τη συνεισφορά τους και για τα έγγραφα μας έχουν στείλει. Ξέρω ότι θα υπάρχουν και ερωτήσεις προς εσάς προς το τέλος. Ερχόμαστε στο τέλος του χρόνου μας που είναι 5.30 και θα δώσω στον εισηγητή την ευκαιρία να έχει τον τελικό λόγο. Απλώς προηγουμένω όμως θα ήθελα να ζητήσω από τον Κλασβίνε να κάνει κάποια σχόλια αν θέλει. Ξέρω ότι είναι πολλά αυτά τα οποία θα μπορούσε να πει, αν μπορούσε μονάχα για ένα-δύο λεπτά να κάνει κάποια σχόλια και μετά μπορούμε να επανέλθουμε στη συνέχεια στα θέματα αυτά. Χαίρομαι που μπορώ να σας δώσω όμως το λόγο για μερικές σκέψεις σε σχέση με αυτά που ακούσατε ήδη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα είμαι σύντομος και θα σταθώ σε ένα-δύο σχόλια. Κάμποση, είπαν εδώ στο πάνελ ότι πρέπει να βασιστούμε στην Γενική Συμφωνία για τους Δημόσιους Διαγωνισμούς και Διεθνή Συμφωνία είναι αυτή για με τρίτες χώρες και να εμπνεύσει την πρότασή μας στη διατύπωση. Εάν δείτε όμω αυτή τη γενική συμφωνία, δεν εκφράζει μόνο γενικές αρχές αλλά και προθεσμίε, ε, κριτήρια επιλογής, ε, αυστηρέ διατάξει. Ε, δεν είναι λοιπόν τόσο απλό. Ε, είναι περισσότερο από αυτό που βλέπει κανεί από πρώτη όψεω. Έπειτα στην οδηγία θέλαμε περισσότερο σε σχέση με την Γενική Συμφωνία. Είναι μια εργαλειοθήκη που πάντοτε είναι ελκυστική. Αλλά εργαλειοθήκη έχουμε και εμεί. Κοινωνικά κριτήρια που δεν υπάρχουν εκεί, περιβαλλοντικά που δεν υπάρχουν, ηλεκτρονικέ διαδικασίε που αναφέρονται ακροφυγώ και την ευκυβερνησία, την σαφήνεια, την καινοτομία όλα αυτά, εάν θέλουμε να υπάρξουν, επειδή δεν είναι μέρη τη Γενική Συμφωνία, θα πρέπει να αναφερόνται στην οδηγία. Θα πρέπει λοιπόν να κάνουμε περισσότερα για τι διαδικασίε και να δώσουμε περισσότερη έμφαση σε ορισμένα χαρακτηριστικά για να καταλήξουμε μια χρήσιμη εργαλειοθήκη. Είναι πολύ εύκολο λοιπόν να λέει κανεί, α πάρουμε τη Γενική Συμφωνία περί δημόσιων διαχωρισμών και να βασιστούμε σε αυτή. Δεν είναι αυτό ο μόνο σκοπό τη οδηγία. Για τα ανώτατα όρια, μια και αναφερθήκατε στη Γενική Συμφωνία, έχει τα όρια παρόμοια αυτά που έχουμε και εμεί στι ισχύουσε οδηγίε. Εάν λοιπόν θέλετε να εμπνευστούμε από τη Γενική Συμφωνία, θα πρέπει να μείνουμε στα ίδια ακριβώ όρια για την επιμνησία. Καταλαβαίνω. Και το έδειξαν και οι διάφορε αναλύσει, ότι πρέπει να δούμε προσεκτικά τι εμπεριέχει η πρόταση. Από την άλλη, όμω, θεωρούμε ότι είναι σημαντικό και δεν είναι θέμα μόνο άχθου, είναι και θέμα τη ιδιοποίηση από τα κράτη-μέλη. Τι όλε διαδικασίε. Δηλαδή οι κανόνε που θα θεσπίσουμε να ισχύουν πραγματικά. Εδώ λοιπόν είναι θέμα διανομή καθηκόντων, κατανομή μάλλον καθηκόντων και θέμα αρχών. Αυτό όμω θα το δούμε, θα το συζητήσουμε, θα το συζητήσει και το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και το καθεξή. Νομίζω λοιπόν ότι είναι σημαντικό γενικώ κάτι να υπάρχει. Να υπάρχει ένα μηχανισμό εξακρίβωση τη ε, συμμόρφωση σε επίπεδο Επιτροπή. Δεν μπορεί να το κάνει αυτό η Επιτροπή με τι ε, διαδικασίε παραβάσει. Τέλο, το θέμα των κοινωνικών υποχρεώσεων αληθεύει ότι κάτι που θα έπρεπε να το δούμε προσεκτικότερα είναι οι υπεργολαβίες και τι υποχρεώσεις προκύπτουν. Για τον ε, βασικό ε, ανάδοχο του έργου, τον πρώτο ανάδοχο του έργου σε σχέση με τους υπεργολάβους. Μπορούμε να εξακριβώσουμε τη συμμόρφωση του ανάδοχου, αλλά θα πρέπει να είναι δυνατό αυτό και για του υπεργολάβους. Θα σταματήσω εδώ γιατί υπάρχουν πάρα πολλά θέματα. Σας ευχαριστούμε. Νομίζω κάποια σημεία τέθηκαν και σε σχέση με την έννοια της καινοτομία. Και αυτό θα πρέπει να το έχουμε υπόψη και να σκεφτούμε αυτά που μας είπε ο κ. Βάης. Κυρίες και κύριοι, τώρα να ευχαριστήσω και τον Μάρκ Ταραμπέλα που διοργάνωσε αυτή την ακρόαση σε συνεργασία με τους κοιόδης εισηγητές. Και Μάρκ, να σου δώσω το λόγο να κάνεις κάποιες καταληκτικές παρατηρήσεις ή να θυμίσεις σε όλους ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα που ακολουθεί. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, αγαπητέ Μάλκομ. Εντάχει, θα αντισταθώ να συμπληρώσω από κύριο Σβίγκλε, διότι δώστε το παράδειγμα του ΠΟΕ, ιδίω ο κύριο Σάρφ. Να πω απλώς ότι εάν κάναμε ό,τι γίνεται στον ΠΟΕ θα μας είχαν απολύσει. Γιατί αν θυμηθούμε τι έγινε στο γύρο της Ντόχα, τα πράγματα δεν πήγαν πολύ καλά. Μάλλον βλάβη είχαμε. Ειδικά εάν δούμε τι έγινε στο γεωργικό τομέα, δεν θα έπαιρνα ποτέ τον ως παράδειγμα. Αλλά να δούμε τι μας απασχολεί σήμερα και τι θα μας απασχολήσει και στο μέλλον επί μακρόν. Η διοργάνωση των δημοσίων διαγωνισμών όπως να την εξετάζει η Επιτροπή από την περασμένο Δεκέμβριο. Αυτό αυτέ ε, οι προτάσει προφανώ προκαλούν επικριτικά σχόλια και είναι λογικό να δοθεί και έμφαση στι αρνητικέ παρατηρήσει. Θα γίνουν προσπάθειε διόρθωση και προσαρμογή, όμω ο βασικό στόχο, όπω έχει τεθεί, όπω έχει δηλωθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον οποίο συμμερίζεται το σύνολο των ε, συμμετεχόντων στην όλη διαδικασία είναι να γίνουν πιο αποτελεσματικέ οι διαδικασίε των δημοσίων διαγωνισμών, θυμίζοντα ότι μιλάμε για το σύνολο των ε, δημοσίων προμηθειών. Όχι μόνο όσων υπόκειται στο ευρωπαϊκό δίκαιο, μιλάμε για ένα συγκεκριμένο ποσοστό του ΑΕΠ. Τα κράτη-μέλη κάποιες φορές ε, μέχρι ένα επίπεδο ε, υπόκεινται στις ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις, αλλά κάποιες φορές οι δραμοδιότητες είναι καθαρά εθνικές. Μιλάμε λοιπόν για το σύνολο των διαγωνισμών. Επίση η αντικατάσταση τη χαμηλότερη τιμή με την έννοια τη προσφορά που οικονομικώ θα είναι πιο λογική, πιο αποφελή. Με κριτήρια ε, κοινωνικά, περιβαλλοντικά, κριτήρια κύκλου ζωή. Όλα αυτά είναι λογικά. Θεωρώ ότι είναι θετικά σημαία. Καταχαιρετίζω. Η απλούσταση τη διαδικασία. Όλοι συμφωνούν εδώ. Απλώ πρέπει να τα καταφέρουμε. Και θα υιοθετήσω εδώ την άποψη που ακούσαμε Μπορεί να μην είμαστε βέβαιοι, αλλά είναι. Η προσπάθεια μετράει. Οι διαδικασίε του Κοινοβουλίου είναι επίση περίπλοκε, δημοκρατικέ βεβαίω. Η Επιτροπή Εσωτερική Αγορά, που είναι καθήλυνα αρμόδια, αλλά υπάρχουν και άλλε 7 επιτροπέ που θα γνωμοδοτήσουν. Με χρονοδιάγραμμα που γνωρίζετε. Πρώτα απ' όλα, τροπολογίε 18 Απριλίου, 8 Μαου με 8 Ιουνίου. Μεγάλο διάστημα για την υποβολή τροπολογιών. Τέλο πάντων, αυτή είναι η ελευθερία που επικρατεί στην ε, κοινοβουλευτική διαδικασία και μετά 7 επιτροπέ θα εξετάζουν το των Τροπολογιών για να καταλήξουμε σε απόφαση στην ε, δική μα επιτροπή στι 10 Οκτωβρίου με ψηφοφορία που μπορεί να μην γίνει και σε αυτή την αίθουσα. Αλλά τέλο στην Ολομέλεια, χωρί να είμαστε βέβαιοι, ψηφοφορία στην Ολομέλεια τον Δεκέμβριο. Γιατί, Γιατί Πρέπει να λάβουμε υπόψη και τι παράλληλε διαβουλεύσει στο Συμβούλιο. Εδώ να χαιρετήσω και την Ιδανική Προεδρία που έχει εγκρίνει μια σαφή μεθοδολογία εργασία με του ε, συνεργατικού σχηματισμού. Και εδώ προσπαθούμε να εμπνευστούμε και εμεί από αυτή τη διαδικασία, να εργαστούμε παρομοίω, ώστε να ε, προχωρούμε παράλληλα με το Συμβούλιο, εμπνεώμενοι από αυτό, χωρί να ξεχνάμε τα όσα συμβαίνουν εκεί και με τις ε, διάφορες μικρές λεπτομέρειες. Είναι λογικό αυτό. Στο Συμβούλιο έχουμε τους εκπροσώπου των κυβερνήσεων. Γνωρίζουν τις καλέ πρακτικές, αυτές ε, τονίζονται ιδιαίτερω, υπογραμμίζονται κάποια εθνικά παραδείγματα. Μπορεί να δημιουργούν προβλήματα στους μεν, όπως η Εθνική Αρχή Ελέγχου, ο άρθρο 84. Εδώ μεταξύ των ε, εκατοντάδων συμμετεχόντων που συνάντησα, ε, αυτό ήταν αποδεκτό από την πλειοψηφία. Θα πρέπει λοιπόν να το αναλύσουμε από νομική σκοπιά, αλλά αφού δούμε τα χαρακτηριστικά τη πρόταση, βλέποντα τι μέρημνε μπορεί να υπάρχουν και α είναι πολλέ, δεν θέλω εδώ να δώσω κάποια φοβερή πρώτη είδηση. Δεν είμαι γνωστό γι' αυτό, αλλά εάν διαγραφόταν το άρθρο 84, εντάξει, εγώ θα μπορούσα να το δεχτώ, όμω θα πρέπει εντωμεταξύ να εξασφαλίσουμε, όπω η οδηγία του 2004, για την καταπολέμηση των στρατιωτικών συνεπειών στις δημόσιου διαγωνισμού, κατά τη διαφθοράς, κατά των κειμένων στους δημόσιου διαγωνισμού. Εδώ θέλουμε να καταπολεμήσουμε ακριβώ αυτά τα κακό κείμενα. Να είμαστε βέβαιοι ότι όλοι οι δημόσιοι διαγωνισμοί υπόκεινται σε μία αρχή σε κάθε κατό μέλο. Ότι υπάρχει έλεγχο. Το είπατε κύριε Δερουά. Θα πρέπει να είναι είτε οικονομικό έλεγχο είτε δικαιοδοσία. Αλλά αυτό γίνεται για την πλειονότητα των ε, δημοσίων διαγωνισμών. Θα, ίσως πρέπει, να, θα πρέπει ίσως να, να διατυπώσουμε την παράγραφα αυτή. Να μετατραπεί το κείμενο της οδηγίας σε κάτι που δεν φοβίζει. Να μην είναι το μεγάλο τέρας, το λόχνες των δημόσιων διαγωνισμών που τρομάζει τον κόσμο αυτό το θέμα της εθνικής αρχής. Πάντω, χωρί να μπω στι λεπτομέρειε του θέματο, θα έχετε δει στο έγγραφο εργασία που σα έστειλα ότι κάποια πράγματα αναφέρονται. Προφανώ, τα κοινωνικά κριτήρια αναφέρονται. Η κυρία Νίλσον μα είπε ότι αν μπορούσαν να γίνονται σεβαστά τα δικαιώματα των εργαζομένων θα ήταν ήδη κάτι. Μπορούμε να πάμε και παραπέρα. Αλήθεια είναι, αλλά ήδη σήμερα γνωρίζουμε ότι εξαιτία ιδιαίτερω τη υπεργολαβία, τη ορευτική υπεργολαβία, τα θεμελιώδη δικαιώματα δεν γίνονται καν σεβαστά. Πολλά χάνονται στο δρόμο, διότι σε κάθε τομέα της, σε κάθε κρίκο της αλυσίδας. Κάποια χρήματα μπαίνουν στην τσέπη, οι επιχειρήσεις δεν σέβονται τίποτα, δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη, μόνο το οικονομικό όφελος υπερισχύει και εις βάρος της αναθέτουσας αρχής του φορολογουμένου και τελικά ποιος καταλήγει να δουλεύει. Μια επιχείρηση που δυστυχώς και αυτό πρέπει κανεί να το καταγγέλει, μια επιχείρηση που υποχρεώνει του εργαζομένου να εργάζονται σε συνθήκε απαράδεκτε για του ευρωπαϊκού κανόνε. Παράνομη λαθρέα εργαζόμενοι που εργάζονται τη νύχτα από έργα που έχουν αντεθεί μέσω δημοσίων διαγωνισμών. Χρόνο. Πω πω, πέντε λεπτά. Τέσσερα είκοσι έχω μιλήσει. Ολοκληρώνω λέγοντας ότι, χωρίς να θυμίσω όλες τις λεπτομέρειες τη σημερινή συζήτηση, ναι, θα συνεργαστώ με του συναδελφού που είναι στι έχουμε ήδη πολύ ενδιαφέρουσε συνομιλίε με την παρουσία του κ. Βίγκλε στο Στρασβούργο και παράλληλα και στι Βρυξέλλε. Θα επαναλάβουμε αυτή την εμπειρία και στην Ολομέλεια του Στρασβούργου. Δεν θα ξεχάσω του ε, συντάκτε νομοδοτήσεων των 7 επιτροπών. Θα κανονίσουμε κοινέ συναντήσει, ώστε να ενημερωνόμαστε αμοιβαίω για τι καλέ πρακτικέ, τι νέε ιδέε που μπορούν να προκύψουν σε επίπεδο επιτροπή, Άρα θα πρέπει να αναζητήσουμε ισορροπία μεταξύ απλούστευση του ε, συμφέροντος των επιχειρήσεων και ιδίως των μικρομεσαίων που θέλουμε καλύτερα και ευκολότερα να συμμετέχουν στις διαδικασίες δημόσιων διαγωνισμών και τέλος των αναθετουσών των αρχών ανάθεσης. Διότι εκείνοι στα χέρια τους τα χρήματα των φορολογουμένων και πρέπει να τα διαθέσουν. Εκεί Εκείνοι αποφασίζουν. Αυτή η μεταρρύθμιση λοιπόν θα πρέπει να είναι προ όφελό του. Διότι διδάλω χάνουμε τελείω το στόχο για τον οποίο εργαζόμαστε. Ευχαριστώ Πρόεδρε και με συγχωρείτε που σα μακρηγόρησα. Well, Χαιρόμαστε για τον ενθουσιασμό σας και τη δέσμευσή σας. Ήταν πάρα πολύ καλά αυτά που ακούσαμε για την αντιμετώπιση σας. Το πιο σημαντικό στοιχείο είναι ότι στις 18 Απριλίου θα στείλετε την έκθεσή σας για μετάφραση. Σας ευχόμαστε καλό Πάσχα <clears throat> καθώς θα δουλεύετε σε αυτό το θέμα. Η επόμενη συνεδρίασή μας λοιπόν θα είναι στις 8 Μαΐου που θα έχουμε την ευκαιρία να επανέλθουμε σε αυτή την έκθεση. Για αυτούς που παρακολουθούν, ίσως θέλετε να τη σημειώσετε, θέλω να ζητήσω σε όλους να χειροκροτήσουν τους, ε, τα μέλη του πάνελ, τους ομιλητές μας για τις θαυμασίες παρουσιάσεις τους. Και έτσι κλείνουμε το δημόσιο τμήμα της συνεδρίας της Επιτροπής. Οι συντονιστές θα πρέπει να συνέλθουν και να συνεδριάσουν σε λίγο. Θα ήθελα να παρακαλέσω λοιπόν όλους και τα μέλη του κοινού <clears throat> να αποχωρήσουν στο εδώ πιο γρήγορα γιατί έχουμε να κάνουμε ένα σημαντικό έργο σε σχέση με τη σχεδιασή του έργου της Επιτροπής στους επόμενους εβδομάδες και μήνες. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας.